Για colleagues, let's start. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας παρακαλώ, καθίστε. Πρώτα απ' όλα. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων Το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται για μια στιγμή κρίσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε έναν συνδυασμό, ε, μια συζήτηση ε, μεταξύ του ε, εθνικού και του ευρωπαϊκού επίπεδου είναι στην κατάλληλη στιγμή καθώς είμαστε τώρα σε μια κάμπη κατά την οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούλιο οι συστάσεις άνα χώρα και τώρα πρέπει να εφαρμοστούν στον εθνικό προϋπολογισμό. Και με τη νέα διαδικασία που προβλέπει έναν πιο έντονο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα Βεβαίως ε, είμαστε στο δεύτερο μισό του χρόνου. Λοιπόν, ε, βλέπετε πως είμαστε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή και η συγητής είναι ο κύριος Ροζάτη, στον οποίο θα δώσω αμέσως το λόγο. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής μας ε, συζήτησης είναι να συνεισφέρουμε στην συζήτηση πριν την επίσημη έγκριση της έκθεσης από το Κοινοβούλιο για να αντιδράσουμε και σε αυτά τα οποία έχει πει η Κομισιόν εντός του 2015 πριν η Κομισιόν δημοσιεύσει την ετήσια έρευνά της για την ανάπτυξη η οποία θα θέτει και τους ε, στόχους τους οικονομικούς αλλά και τους δημοσιονομικούς για το επόμενο έτος. Δεδομένου δε του σημαντικού αριθμού βουλευτών θα δώσουμε πρώτα απ' όλα τον λόγο σε εθνικούς βουλευτές και βεβαίως ε, θα προσπαθήσουμε όλας ε, να δώσουμε τον λόγο και σε ευρωβουλευτή από την ίδια χώρα. Θα χρησιμοποιούμε λοιπόν μια κάρτα για να διευκολύνουμε την συζήτηση. Αν ευρωβουλευτές ή οι βουλευτές ε, θέλουν να μιλήσουν μπορούν να δώσουν την κάρτα στον κλητήρα. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση. Ο κύριος Ροζάτη έχει το λόγο για να παρουσιάσει την έκθεσή του για 10 λεπτά. Δαρίε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να εκφράσω πρώτα απ' όλα την ε, ικανοποίησή μου για την ευκαιρία που έχουμε να συναντηθούμε εδώ πέρα με βουλευτές από τα κράτη-μέλη και να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό κομμάτι του Ευρωπαϊκού Εξαμένου που είναι ένας βασικός μηχανισμός για να συντονίζουμε τις ε, οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Η έκθεση αυτή την οποία αναφέρατε κύριε Πρόεδρε αναφέρεται σε μια σειρά εγγράφων που προετοίμασε η Κομισιόν και το Συμβούλιο ξεκινώντας από την ετήσια έκθεση ανάπτυξης ε, πέρσι τον Δεκέμβριο ένα έγγραφο δηλαδή το οποίο θέτει το πλαίσιο για να προετοιμάσουμε τις ε, συστάσεις. Αναχώρα με βάση λοιπόν αυτή την έρευνα, την ετήσια για την ανάπτυξη, η Κομισιόν προετοιμάζει εθνικές εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τα εθνικά προγράμματα σταθερότητας ε, και σύγκλησης. Και βεβαίως, επί τη βάση των πληροφοριών που στέλνουν τα κράτη-μέλη, η Κομισιόν προετοιμάζει συστάσεις ε, προς το Συμβούλιο. Όπω είπαμε, η Κομισιόν ε, έλαβε αποφάσεις στις ε, συστάσεις ε, αναχώρα φέτος. Είπατε λοιπόν πως αποτελεί μέλος του ετήσιου κύκλου τη σημερινή συνεδρίαση και ακριβώ έχει στόχο να αξιολογήσει τις συστάσεις αναχώρας Κομισιόν όπως τις προετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση και την απόφαση του Συμβουλίου του Ιουλίου. Ο γενικότερος στόχος των συστάσεων είναι να δώσει στα κράτη-μέλη κάποιες σύμβουλες και κάποιες συστάσεις για το πώς θα διαμορφώσουν την εθνική οικονομική πολιτική για να ανταποκριθούν στις πιο σημαντικές προκλήσεις ε, και να εφαρμόσουν ε, τις ε, πιο σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ακολουθούνται οι προτεραιότητες όπως έχουν καθοριστεί στην ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη. Οι συστάσεις αναφέρονται σε δύο τομείς ε, βασικά. Ο πρώτος τομέας είναι δημοσιονομική και φορολογική πολιτική που θα πρέπει να σέβεται το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης ε, και το διπλό και το εξαπλό πακέτο και ο δεύτερος τομέας είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών και να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους όπως αυτοί αναφέρονται στην στρατηγική 2020. Φέτος οι συστάσεις να αντικατοπτρίζουν ε, τις ε, παλαιότερες αξιολογήσεις που είχαμε κάνει και έχουν ε, βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να αναφέρω δύο σημαντικές βελτιώσεις στις φετινές συστάσεις. Πρώτον, δημοσιεύτηκαν πολύ νωρίτερα φέτος. Τρεις μήνες νωρίτερα. Και βεβαίω το σκεπτικό εδώ πέρα είναι να δοθεί περισσότερο χρόνο στα κράτη-μέλη και ειδικά στα κοινοβούλια να συζητήσουν τα σχέδια ε, συστάσεων, να τα αναλύσουν εις βάθος ε, και να καταλήξουν σε αποφάσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την εφαρμογή τους. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή φέτος είναι πως ε, οι συστάσεις είναι πολύ πιο στοχευμένες ε, σε βασικές προτεραιότητες. Η Κομισιόν έχει καταβάλει προσπάθειες ε, να αποφύγει την διατύπωση ευρύτατων στόχων. Ανταυτού εστιάζει σε βασικές προτεραιότητες. Και η νέα αυτή προσέγγιση είναι μια προσέγγιση με την οποία συμφωνεί το Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε δηλαδή με τις στάσεις της Κομισιόν σε αρκετές στοιχές. Πρώτα απ' όλα συμφωνούμε με την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε κάποια σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, αλλά συμφωνούμε πως τα θεμέλια αυτής της ανάκαμψης είναι ακόμα εύθραυστα και πρέπει να γίνουν ε, πολύ περισσότερα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψει σε έναν δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το να εστιάσουμε σε τέσσερις προτεραιότητες κλειδιά, δηλαδή αύξηση των επενδύσεων, μια δημοσιονομική εξυγίανση φιλική προς την ανάπτυξη, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και βεβαίω κάποιες πολιτικές ε, προσανατολισμένες προς το μέλλον. Επίσης, συμφωνούμε με την Κομισιόν πως μέχρι στιγμής ε, η εφαρμογή των συστάσεων από τα κράτη-μέλη δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Μπορούμε να μιλήσουμε μάλιστα για κακή εφαρμογή, μέτρια. Και θα έλεγα πως ένα 10% έχει εφαρμοστεί πλήρως και άλλο ένα 10-15% εν μέρη από τις συστάσεις. Οπότε θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων από τα Εθνικά Κοινοβούλια για το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί το ποσοστό εφαρμογής. Επίσης, συμφωνούμε με την Κομισιόν πως χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην έκθεσή μα αναφέρουμε συγκεκριμένου τομεί όπου πρέπει να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μεταρρυθμίσεις ε, στην αγορά εργασίας, ε, στην ε, λειτουργία της ενίας αγοράς, το να μην υπάρχουν δηλαδή εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, διαστατικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημοσίων οικονομικών, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα εθνικά τα ταμεία, για να αναφέρω τα σημαντικότερα μόνο. Βεβαίως, ε, ακομα ακόμα κάποια κράτη-μέλη έχουν πολλά, πολύ μεγάλα υπερβολικά επίπεδα δημοσίου χρέους. Ε, συνιστούμε πιο ενεργή δημοσιονομική πολιτική και μάλιστα ε, να χρησιμοποιηθεί αυτή με τρόπο αντικυκλικό στις ε, χώρες εκείνες οι οποίες έχουν κάποιο περιθώριο και των οποίων το επίπεδο χρέους είναι κάτω από το όριο του 60%. Οπότε, όταν μιλάμε για την εξυγίανση των ε, δημοσίων οικονομικών, οι συστάσεις ε, διαφέρουν. Όπως άλλωστε διαφέρει και η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Όταν μιλάμε τώρα για τις ε, συστάσεις, δεν θα τις αναφέρω όλες. Δύο μόνο από αυτές. Ε, μιλάμε για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα κίνητρο και για ιδιωτικά κεφάλαια να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις και ο δεύτερο τομέας είναι το νομικό και θεσμικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και εδώ πέρα ζητάμε από τα κρατη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα τέτοιο περιβάλλον και να δημιουργήσουν συνθήκες οι οποίες θα ευνοούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τις δουλειές. Τέλος. Τέλος, ναι, έχετε 30 δευτερόλεπτα, λέει ο πρόεδρος. Τέλος, μιλάμε για την ε, μέτρια ως κακή εφαρμογή των συστάσεων στα κράτη-μέλη και θεωρούμε πως ένας από τους λόγους πίσω από αυτό είναι η ανεπαρκής ε, εγκόλπωσή τους από τα κράτη-μέλη. Και εδώ πέρα ακριβώς θα θέλαμε μία συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Τέλεια εξηγώ στους ε, φίλους μας ότι έχουμε πλέον νέο κανονισμό και έχουμε ευελιξία στο Συμβούλιο στο Σύμφωνο με συγχωρείτε σταθερότητας και ανάπτυξης αλλά όχι στο χρόνο μιλίας. Οπότε ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά γιατί θα κόβω το μικρόφωνο κατευθείαν. Λοιπόν, για πέντε λεπτά το πολύ και για τον Ευρωβουλευτή και για τους Εθνικούς Βουλευτές. Λοιπόν, ο πρώτος ομιλητής είναι ο Αλφρεντ Σάντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρόλο που κάποιοι βιομηχανικοί δείκτες πρόσφατα ήταν καλύτεροι στην Ευρωζώνη, η ανάκαμψη είναι πολύ εύθραυστη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο υποτίθεται ότι θα συντονίσει τις οικονομικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη για να ενισχύσει την ανάπτυξη. Στο ίδιο έχει δοθεί έμφαση στο πρόγραμμα για το 2015 με τη δημοσίευση των συστάσεων της Κομισιόν για τα κράτη-μέλη το περασμένο Μάιο. Η Κομισιόν θέλει να ευθυγραμμίσει τη διαδικασία σύμφωνα με τις οποίες διατυπώνονται και εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τα κράτη-μέλη. Ε, το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι οι συστάσεις ή δεν εφαρμόζονται καθόλου ή εφαρμόζονται άκαμπτα. Και ένας από τους λόγους είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια δεν αναλαμβάνουν την ιδιοκτησία των ε, ειδικών συστάσεων αναχώρα. Ένα άλλος λόγος είναι ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο υπάρχει στρατηγική πίσω από τις εκάστοτε συστάσεις για την εκάστοτε χώρα, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό, τους, σύνολό ή για την ενίσχυση της συγκεκριμένης χώρας. Άρα έχει έρθει η στιγμή να αξιολογήσουμε κριτικά τον αντίκτυπο και το περιεχόμενο των συστάσεων της Κομισιόν αναχώρα για να γίνουν πιο αποτελεσματικές και να είναι αποδεκτές ως εργαλείο πολιτικής. Και αυτό είναι αναγκαίο, διότι τα αποτελέσματα από πλευράς ανάπτυξης δεν ήταν ικανοποιητικά μέχρι σήμερα και άλλωστε δεν είναι πάντοτε αξιόπιστα τα στοιχεία στα οποία βασίζονται. Για παράδειγμα, Συχνά οι συστάσεις αναχώρα βασίζονται στην υπεραπλουστευμένη άποψη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν μηχανικό και αυτόματο αντίκτυπο στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Και έτσι δηλαδή αν ταυτοχρόνως όλες οι χώρες μεταρρυθμίσουν τις αγορές εργασίας, τότε η έξτρα ζήτηση που θα δημιουργηθεί από τις νέες θέσεις απασχόλησης θα έχει ένα spillover effect, ένα αποτέλεσμα διάδοσης και επέκτασης στο σύνολο της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι εσφαλμένο. Οι κοινωνικές συνέπειες των συστάσεων έχουν αγνοηθεί στην πράξη, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες απότυχαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα της απασχόλησης σε πολλές χώρες. Αν το μεταξύ, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας έχουν διαβρώσει τα εργασιακά δικαιώματα και έχουν ενθαρρύνει την αβέβαιη απασχόληση, την επισφαλή σε όλη την Ευρώπη. Και δεν ε, μπορεί να είναι η πρώτη διαρθρωτική μεταρρύθμιση αυτή της αγοράς εργασίας. Αντιθέτως πρέπει να αναδείξουμε τα κρυφά μονοπόλια, την ε, ε, καταπολέμηση αυτών της ε, κρατικής γραφειοκρατίας, τον εξυγχρονισμό του δικαιακού νομικού συστήματος. Αυτά να έχουν την πρωτοκαθεδρία από πλευράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεις. Από πλευράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι αποκλήσεις οξύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση που έχει ως βασικό στόχο τη σύγκληση. Δεν έχουμε τα εργαλεία που θα αντισταθμίσουν το όλο και μεγαλύτερο το χάσμα που παρατηρείται μεταξύ Βορρά και νότο, Νότου. Ε, είναι αντιπαρηγωγικό να έχουμε περισσότερη Ευρώπη όταν δεν έχουμε πολιτική που εντάσσουν τις συστάσεις άνα χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με στόχο την μείωση των ανισοτήτων και την αύξηση της σύγκλησης. Και έτσι θα ήταν πιο εύκολο αν αυτό υπήρχε πράγματι τα κοινοβούλια να αναλάβουν την ιδιοκτησία των συστάσεων που προτείνονται αναχώρα. Ευχαριστώ. Στάνισλαφ Πόζοκ. Παρακαλώ. Από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το CSR country-specific recommendations, τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα. Εξέτασα την, μελέτησα την έκθεση και αναρωτήθηκα το εξής. Ε, με ποια βάση γίνεται η δουλειά για τα εκάστοτε κράτη-μέλη Κοιτάζω το πίνακα των συστάσεων και θέλω να σας προβάλλω το παράδειγμα της ε, Πολωνίας. Έχουμε στοιχεία για αυτά που έχουν εφαρμοστεί, για, το, αυτά που δεν έχουν εφαρμοστεί, για το ποια ακριβώς ήταν η πρόοδος, αν έχει υπάρξει τελικά. Ποιος είναι ο αποφασιστικός παράγοντας του εθνικού επίπεδου που μετράει στην εφαρμογή ή στη μη εφαρμογή της χ υψη σύστασης. Ε, για παράδειγμα, η Πολωνία δεν έχει σημειώσει πρόοδο στη σύσταση της εξάλληψης του υπερβάλλοντος αριθμού των συμβάσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Μπορεί αυτό να εξηγηθεί από την οικονομική κατάσταση της Πολωνίας. Αναρωτιέμαι, πώς παίρνουν τις αποφάσεις τα κράτη-μέλη και σε ποιο βαθμό οι κυβερνήσεις αισθάνονται υπεύθυνε για την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Και αυτές οι συστάσεις φαίνονται δεσμευτικές, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φαίνεται ότι ο νέος κανόνας για το χρόνο ομιλίας έχει ε, ως αντίκτυπο τον αυτοπεριορισμό των μελών ακόμα ε, και σε πιο σφιχτά περιθώρια από αυτά που τους δίνουμε. Από πλευράς Άλτε, ο κύριος Νίλς Άστρομ που είναι δεν είναι εδώ προχωρούμε δεν ξέρω αν το βλέπετε είναι εδώ Εσείς παίρνετε το λόγο εξ ονόματος του Γάλντε. Σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Ντεμάζη. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Έχω μελετήσει την έκθεση αυτή. Όπως ξέρετε η προσέγγιση μας είναι αρκετά κριτική. Δεν συμφωνούμε με τη θετική ε, προοπτική της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ η κίνδυνη. Άλλωστε η Τράπεζα για τη Διεθνή Επίλυση των Διαφωνιών έχει ανακοινώσει τις ε, ανησυχίες της. Υπάρχει ερώτηση γιατί η απόδοση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αδύναμη και ασθενής λόγω της λιτότητας και των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Υπάρχουν οι προσδοκίες ότι η τελευταία δέσμη μέτρων που έχει συμφωνηθεί με την Ελλάδα θα ενισχύσει την ύφεση Πολλοί το περιμένουν αυτό και συμφωνούμε. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ασκούν πίεση ε, στα ημερομίσθια, στις συντάξεις. Όλα αυτά πλήττουν την εσωτερική ζήτηση και άρα υπονομεύουν ακόμα περισσότερο το δρόμο της Ευρώπης προς την οικονομική ανάκαμψη. Πάρα πολλές είναι οι ανεπάρκειες και λήψει της έκθεσης σε σχέση με ε, τη δουλειά του Eurogroup. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση έκανε η νομική υπηρεσία ε, της Deutsche Bank, Deutsche Bank και ε, εμφανίστηκε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει πρωτόκολλο το Eurogroup, δεν έχει διαφάνεια, δεν έχει δημοκρατική νομιμότητα, επομένως ενδεχομένως δεν έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις που πήρε τους τελευταίους μήνες. Οι διαδικασίες μακροοικονομικών ισορροπιών θα πρέπει να εκφράζουν και το πρόβλημα των μεγάλων εξαγωγικών πλεονασμάτων ορισμένων χωρών, ε, οι οποίες ε, δεν τιμωρούνται, ενώ τιμωρούνται τα υπερβολικά ελλείμματα άλλων χωρών. Ίσως τελικά η Γερμανία πρέπει να κάνει περισσότερο για να ενισχύσει την εσωτερική της ζήτηση και συστηματικά παραμερίζεται η υπερβολική συγκέντρωση του ε, κρατικού χρέους. Η Ισπανία και η Ιρλανδία έχουν υποφέρει από αυτό. Και άλλωστε η έλλειψη ροών στην πίστη, στην πίστοση, οφείλεται στην λιτότητα. Υπάρχει έλλειψη επενδύσεων, δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πραγματικά δημόσιο κρατικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο θα ενισχύσει τη ζήτηση. Και το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνει συνταγές που δεν έχουν δουλέψει στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να αποδώσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πρώτος ομιλητής, Herbert Hirte, από τη Γερμανική Bundestag. Για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε να πω λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρώτα απ' όλα ήθελα να εκφράσω την άποψη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της ε, συμπολίτευσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι σωστή προσέγγιση γιατί συνεισφέρει και στην ε, δημοσιονομική εξυγένση ακόμα και σε άλλες ε, χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε τα προγράμματα επενδύσεων, ευχαρίστως. Αλλά τα χρέη θα πρέπει να βρίσκονται σε μία αναλογία με τις βιώσιμες επενδύσεις. Τα χρέη και σε καιρούς ε, καλούς ε, είναι μία προσέγγιση η οποία δεν είναι σωστή. Επίσης, με μεγάλη ανησυχία διαπιστώνουμε πως δεν εξετάζονται επαρκώς οι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεν είναι πλήρης οι αναλύσεις της Eurostat και πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Το τρίτο που αφορά την εξυγίανση των προπολογισμών και αναφέρθηκε ήδη είναι το ότι αφενός θα πρέπει να υπάρξει κάποια ελάφρυνση του χρέους αλλιώς είναι αναπόφευκτη μια έξοδος από την Ευρωζώνη. Εμείς ε, είμαστε της άποψης πως μπορεί να συνεχιστεί η ένταξη στο ευρώ αρκεί να υπάρχει μια σωστή πολιτική απάντηση σε μια λανθασμένη κατάσταση και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εισαγωγής μιας διαδικασίας κρατικής χρεοκοπίας όπως έχει προτείνει και ο Υπουργός των Οικονομικών μας. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένα τις συστάσεις για τη Γερμανία, παρατηρούμε με ανησυχία την κριτική στο γερμανικό εμπορικό ισοζύγιο και το πλεόνασμά του, που είναι θέμα επιτυχίας ε, οι εξαγωγές και πραγματικά με δυσαρέσκεια σημειώνουν οι Γερμανοί πως η επιτυχία πλέον θεωρείται κάτι το αρνητικό από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, εντάξει, είναι κατανοητά τα επιχειρήματα, αλλά πολιτικά ε, δεν το βρίσκουμε πάρα πολύ εύστοχο. Και τέλος, υπόθηκε ήδη πως η δημοκρατική νομιμοποίηση της ε, Ευρωζώνης ε, δεν είναι επαρκής ε, και αυτό μάλιστα ήταν η άποψη της νομικής υπηρεσίας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής αλλά δεν είναι η θέση της Ολομέλειας του σώματος. Αυτό θέλω να το τονίσω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας κάνω μια ερώτηση επί τη ευκαιρία. Γιατί Βεβαίως ε, δεν είναι θέμα κριτικής, αλλά υπάρχει ένα όριο για το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου. Ε, ποια είναι η άποψή για αυτό το στοιχείο συγκεκριμένα. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση. Η ερώτηση αφορά... Ε, ναι, πράγματι συμφωνώ. Δεν είναι δυνατόν να ασκούμε κριτική σε ένα κράτος μέλος επειδή εξάγει. Αλλά σύμφωνα με τους ε, κανόνες που έχουμε στο, στο σύμφωνο σταθερότητας ε, υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο θεωρούμε πως και το πλεόνασμα είναι μια μακροοικονομική ανισορροπία. Τι θα απαντούσατε σε αυτό. Μια αυτό ανέφερα ακριβώς. Ότι αντιλαμβανόμαστε την συνολική άποψη της Κομισιόν και μας είναι γνωστή. Απλά σας λέω πως είναι κάτι το ψυχολογικό, δηλαδή ότι ασκείται κριτική στην εξαγωγική οικονομία, γνωρίζοντας βεβαίως ότι αυτή η εικόνα μπορεί από ευρωπαϊκή σκοπιά να θεωρηθεί αρνητική το αποτέλεσμα που έχει αυτό στην Γερμανία και αυτό είναι μια ανησυχία πολιτικά είναι κάτι το αρνητικό. Γιατί τι γίνεται ουσιαστικά εδώ πέρα ασκούμε μια κριτική σε ένα επιτυχημένο σύστημα. Ευχαριστώ. Μάρκο Βάλι είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Παρεμβαίνω ως σκιώδης ε, εισηγητής για την ομάδα μου, την FDD. Ε, εγώ αμέσω ε, θα αναφερθώ στο θέμα του γερμανικού πλεονάσματος γιατί είναι κρίσιμο αυτό και έχει αναφερθεί και στην έκθεση Μπερές αλλά και σε προηγούμενα κείμενα που αφορούσαν τις ε, διαδικασίες και τις συστάσεις ανακράτως για κάθε εξάμεινο πέρυσι. Ε, πρόκειται για έναν κανόνα ο οποίος θα έπρεπε να εφαρμόζεται, όμως όταν τα συμφέροντα του μεγαλύτερου μετόχου της Ευρώπης ε, γίνονται, μπαίνουν στο στόχαστρο των κανόνων, τότε πια οι κανόνες ε, λέμε δεν είναι σωστοί. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε γιατί δεν ενεργεί η Κομισιόν, γιατί αυτή η έλλειψη ισορροπίας αφορά ολόκληρη τη συζήτηση για την ΟΝΕ. Δηλαδή, η Ευρωζώνη υποφέρει ε, από διάφορα σκάνδαλα, όπως το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία που υιοθετούν ειδικά προνομιακά προλογικά καθεστώτα. Ε, η Γερμανία έχει υπερβολικό πλεόνασμα. Μπορεί δηλαδή να υπάρξει μια κατάρρευση. Και το είπε και ο Γιούνκερ, ότι δηλαδή στην Ένωση δεν υπάρχει Ένωση. Την Τετάρτη το είπε μόλις ο Γιούνκερ. Ε. Σε αυτό το απόλυτο τέλμα προχωρούν λοιπόν και άλλες ιδέες για να προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει ε, για την εργασία και να μπορέσουμε κάπως να φέρουμε την πολιτική κατάσταση των χωρών σε μια πιο νυφάλια κατάσταση. Τώρα πιο συγκεκριμένα, πέρα από την, από την υπογράμμιση αυτών των ε, της ατυπικής συμπεριφοράς της Κομισιόν απέναντι στη Γερμανία και έπειτα και στην Ολλανδία ε, το θέμα της ευελιξίας εντάξει, αλλά θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χώρος στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστές πολιτικές ε, για να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα απασχόλησης. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια ε, ευρωπαϊκή πολιτική και όχι απλώς μια πολιτική περιορισμού του πληθωρισμού. Επίσης, ε, είμαστε κατά των ε, του άγριου φιλελευθερισμού που υποστηρίζουν τα λόμπι, αλλά θέλουμε πολύ περισσότερο να υπάρχουν προβλέψεις κοινωνικού τύπου, γιατί είδαμε στην Ελλάδα τι γίνεται. Πολύ, πολύ μεγάλη φτώχεια, καταστάσεις όπου η λιτότητα τελικά έχει αποδειχθεί ακόμα πιο ζημιογόνα για τον ίδιο τον πληθυσμό. Με αποτέλεσμα την ε, άνοδο ακραίων δυνάμεων. Είναι σημαντικό λοιπόν κατά τη γνώμη μου για να συζητήσουμε μαζί για να καταλάβουμε ποια ακριβώς είναι η κατάσταση αυτής της νομισματικής ένωσης με όλα τα κρατημέλη, να δούμε μήπως θέλουμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουμε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρώπη που να βασίζεται σε ένα σωρό παράδοξα ε, ε, και να δούμε πώς θα πρέπει να χειριστούμε την αναπτυξιακή πολιτική, τις περιφερειακές πολιτικές όπου υπάρχουν διάφορα συμφέροντα στο προϋπολογισμό, να δούμε πώς θα μπορέσει να προχωρήσει η Ευρώπη και μετά βέβαια οι ίδιοι εκλογείς θα κρίνουν το τι έχουμε κάνει. Ευχαριστώ. Η Μπάρμπαρα Κάπελα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε πως το 2014 Μόλις 12% των στάσεων εφαρμόστηκαν πλήρως και ένα 10 με 15% εν μέρη. Μιλάμε δηλαδή για ένα 25% το πολύ ποσοστό εφαρμογής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούν να ανέβουν αυτά τα νούμερα. Η λίστα μπορούσε να είναι η ένταση του ρόλου των εθνικών ε, κοινοβουλίων ε, στην διαδικασία αυτή. Θεωρώ έτσι πως θα αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης τα κράτη-μέλη. Γιατί αυτό βεβαίως μετά οδηγεί και σε μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμογής. Αλλά ας μην είμαστε αφελείς. Το θέμα δεν είναι ότι δεν θέλουν να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη τις μεταρρυθμίσεις, αλλά υπάρχουν πολιτικά εμπόδια, εκλογές. Είναι αργά σε μια θητεία και είναι δύσκολο να κάνουν κάποιες οδυνηρές μεταρρυθμίσεις. Οπότε χρειαζόμαστε πράγματι ανάπτυξη, απασχόληση, γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εδώ πέρα ακριβώς ε, πηγαίνουν οι συστάσεις αυτές και το εξαπλό και το διπλό πακέτο. Εάν τα καταφέρουμε λοιπόν, εάν καταφέρει η Ευρώπη να τα εφαρμόσει αυτά, θα αποκτήσει ξανά ανταγωνιστικότητα. Σημαντικό αυτό λοιπόν το οποίο είπε ο εισηγητής, ειδικά για τα κράτη-μέλη που είναι εδώ πέρα σήμερα. Το ότι δημοσιεύτηκαν δηλαδή νωρίτερα οι συστάσεις και ότι είναι εστιασμένες στη δημοσιονομική πειθαρχία, την απασχόληση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θεωρώ πως έτσι θα καταφέρουμε να αξιθεί ο βαθμός ε, το ποσοστό εφαρμογής. Και ελπίζω να καταλήξουμε, όπως είπα, σύντομα στα εθνικά σχέδια δράσης. Thank you. Now go back to national parliaments. Uh, Katri Kulmini, if I read correctly the name, sorry if I didn't. Uh. Τώρα στα Εθνικά Κοινοβούλια η Κάτρι Κουλμίνη, ζητώ συγγνώμη αν δεν ε, προφέρω σωστά το όνομά σας, από το Κοινοβούλιο της Φιλανδίας. Πρόεδρε, οι κατευθυντηρίες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, καλούν ε, τη χώρα να, έχουμε, να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και να βελτιώσει τη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική στη Φιλανδία. Αυτά ισχύουν για την ε, άρτη εκλεγής κυβέρνηση της Φιλανδίας η οποία εξελέγει τον Απρίλιο. Το ίδιο πιστεύει και εκείνη. Έχουμε έλλειμμα στον προπολογισμό σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάφορα άλλα ζητήματα αντιμετωπίζουμε. Ε, επομένως αναλάβαμε δράση και αυτή η δράση θα μας καθοδηγεί για την επόμενη τετραετία. Είναι σημαντικές οι πολιτικές μας ε, για το ε, σύστημα ασφαλίσεων και το σύστημα κοινωνικής προόνοιας και πρέπει να κάνουμε περικοπές ύψους 4 δις. Αυτό είναι πάρα πολύ για τον προπολογισμό μιας μικρής χώρας όπως η δική μας μέσα σε 4 χρόνια. Και το 2021 ε, το χρέος μας θα αρχίσει να μειώνεται και ε, μέχρι το 2030 θα είναι κατά 10 δις λιγότερο από ό,τι είναι σήμερα. Η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης θα φέρουν αποτελέσματα. Όμως δεν αρκούν οι περικοπές. Σε όλη την Ευρώπη και στη δική μας χώρα χρειαζόμαστε νέες επενδύσεις πάνω σε βασικά έργα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση, με την ψηφιοποίηση, με την βιοοικονομία. Και καταβάλαμε πολλές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση στην Φιλανδία. Σε ό,τι αφορά στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη χώρα μας, να σας πω ότι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα που συζητείται ε, πολύ ε, στη Φιλανδία αυτή τη στιγμή είναι η μεταρρύθμιση του συνδιοξιδιωτικού και η μεταρρύθμιση βασικών πτυχών της αγοράς εργασίας. Όλα αυτά δρομολογούνται, είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση για την Ευρώπη. Η κρίση στην Ευρώπη του καλοκαιριού έδειξε ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Εμείς δεσμευτήκαμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά και ε, μάθαμε, αντλήσαμε διδάγματα από τις συστάσεις της Επιτροπής και ε, ολοκληρώσαμε και χαράξαμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα αναλόγως και αντιστοίχως. Όμως είναι δύσκολο καιρή και είναι δύσκολο να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. You have more time. Ευχαριστώ. Έχουμε και περισσότερο χρόνο αν θέλετε να ε, επεκταθείτε, αγαπητοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου της Φιλανδίας. Παύλο Κουαλιέρη από την Ιταλική Γερουσία, παρακαλώ. Yes. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πιστώνουμε μια θετική αλλαγή στη διατύπωση των συστάσεων αναχώρα, αλλά και στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχουν γίνει κάποιες θετικέ ε, βελτιώσεις. Όμως ταυτόχρονα πιστεύω πως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια αδύναμα σημεία και κάποιες ακόμα σημαντικές βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα να σας δώσω αυτό το γενικό παράδειγμα για το γεγονός ότι αρκετέ συστάσει που σχετίζονται με την Ευρωζώνη αλλά και με την Ευρώπη ολόκληρη δεν αντικατοπτρίζονται στις αναχώρα συστάσεις. Δηλαδή, πρόκειται για συστημικές πολιτικές και αλλαγές που χρειάζονται στην Ευρωζώνη εν γέννη και ε, αυτές οι συστημικές παρεμβάσεις δεν αντικατοπτρίζονται στη συνέχεια στο τι θα πρέπει να επιδιώξει κάθε χώρα και σας δίνω αυτά τα δύο παραδείγματα που έχουν ήδη αναφερθεί σε άλλες παρεμβάσεις. Καταρχήν, πολύ σημαντική προσαρμογή ανάμεσα στις χώρες ε, τις πλανασματικές και τις ελληματικές. Αυτό δεν είναι ίσω σημασία, αντιθέτως είναι πολύ σημαντικό για τη συμπεριφορά της ζήτηση στην Ευρωζώνη εν γέννη και ευρύτερα στην Ευρώπη. Αν δούμε αυτού του είδους τη σύσταση, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αόριστη ανάθεση ε, στις χώρες, ιδιαίτερα για τις χώρες ε, τις πλεονασματικές και από αυτή την άποψη δεν, δεν δίνεται έμφαση σε αυτού του είδους την συμμετρική προσαρμογή. Και αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για την ανταγωνιστικότητα στις τιμές, δηλαδή για να γίνουν προσαρμογές στην ανταγωνιστικότητα των τιμών, αλλά όπως γνωρίζουμε είναι και πάρα πολύ σημαντικό για την ε, βιωσιμότητα του χρέους είναι δηλαδή εξαιρετικά σημαντικό εφόσον θέλουμε να έχουμε ε, βιωσιμότητα χρέους και να έχουμε τη δυνατότητα να γίνουν προσαρμογές ε, που δεν θα είναι πολύ χαμηλά στον πληθωρισμό για τις πλανεσματικές χώρες. Ε, ένα άλλο παράδειγμα είναι η δημοσιονομική στάση, δηλαδή η δημοσιονομική πολιτική για την Ευρωζώνη και για ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια θα ήταν η καλύτερη δυνατή δημοσιονομική στάση η, η βέλτιστη αναφέρεται η ουδετερότητα φέτος και εντάξει αυτό είναι ένα βήμα μπροστά γιατί η ουδετερότητα σημαίνει πως τουλάχιστον δεν είμαστε στις περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές του παρελθόντος. Ωστόσο, ουδετερότητα ε, δεν ορίζεται στις υποδείξεις προς κάθε χώρα. Συμμετρική προσαρμογή λοιπόν και δημοσιονομική στάση. Εκεί θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα ε, ώστε να υπάρχει σχέση ανάμεσα στο ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι της Ευρωζώνης και ποιοι είναι οι υποδείξεις ανά κάθε χώρα. Αυτό έχει σημασία γιατί ε, επηρεάζει την εθνική οικονομία. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αρκετή ζήτηση ε, στην Ευρωζώνη και σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό όλο το σοδυνητικό χώρος να χρησιμοποιείται, να αξιοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Δίνω το παράδειγμα της χώρας μου, γιατί είναι πολύ πιθανό η χώρα μου να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Όχι 0,7% αλλά Μάλλον θα φτάσουμε φέτος 0,9% και ίσως και 1%. 1,6 συγγνώμη του χρόνου. Γιατί, γιατί για πρώτη φορά, λόγω, χάρη στην ευελιξία, μπορέσαμε να έχουμε κάποιο είδου ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το χρόνο. γιατί έχουμε προχωρήσει σε τόσε μεταρρυθμίσεις, έχουμε επενδυτικό προγραμματισμό και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την ίδια ευκαιρία, δηλαδή τη δυνατότητα να έχουμε συνδυασμό μεταρρυθμίσεων επενδύσεων από τη μια πλευρά και ευελιξία από την άλλη. Αυτή η σχέση ανάμεσα στον εθνικό εξωτερική ε, πολιτική και την ευρωπαϊκή εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική και μπορούμε να τη βελτιώσουμε αν θέλουμε να έχουμε καλύτερη συσχέτιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντουάρντο Καπρίτα από την Πορτογαλία. Καλησπέρα σας. Εμείς από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι αυτές οι συναντήσεις διαλόγου ανάμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά την συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής συμβάλλουν καθοριστικά στην εμβάθυνση ενός στρατηγικού συντονισμού ανάμεσα στα κράτη της Ευρωζώνης με την, ε, με την δημοσιονομική εξηγήνση, με την στρατηγική ανάπτυξη ε, και απασχόληση μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύη, στον ευρωπαϊκό χώρο. Γι' αυτό και ακριβώς το Εθνικό μας Κοινοβούλιο που δίδουμε τεράστια σημασία στα τις συζητήσεις που είχαμε φέτος τόσο με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης όσο και με τον Επίτροπο Μοσχοβησή την Επιτροπή Οικονομίας και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μας επισκέφθηκαν. Ε, η, το θέμα είναι ο περιορισμένος χαρακτήρας της συζήτηση ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το, και το Ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να ενισχυθεί η επαφή αυτή και δεν μπορεί να περιορίζεται σε δύο ετήσιες συναντήσεις ε, γιατί κατά τη διάρκεια δύο ώρων στην ουσία παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση πρόοδου. Ωστόσο είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη αυτής της αλλαγής της προτεραιότητας του σχέδιου Juncker στις επενδύσεις. Επίσης ε, η ε, στάση της Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και η πορεία που έχει γίνει προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ευελιξίας από πλευρά της Κομισιόν όσον αφορά την ερμηνεία των κανόνων ε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Γιατί μόνο έτσι είναι δυνατόν να ξεπεραστεί αυτό που είναι ο πολύ αρνητικός ισολογισμός των στρατηγικών προσαρμογής. Η Πορτογαλία ήταν υποκείμενο ε, ενό προγράμματος προσαρμογής στη διάρκεια τριών ετών και ε, αυτό οδήγησε σε πολύ μεγαλύτερη ύφεση από αυτή που είχε προβλεφθεί, επίπεδα ανεργίας ε, πολύ μεγαλύτερα από τα αρχικά προβλεπόμενα, επενδύσεις που ήταν σε επίπεδα αντίστοιχα τόσο μιλώ για το δημόσιες αλλά και για τις ιδιωτικέ επενδύσεις, ήταν τα χαμηλότερα από τότε που μπήκε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίπεδα μετανάστευσης εξαιρετικά ψηλά που ποτέ δεν είχαμε γνωρίσει σε περίοδο δημοκρατίας. Είχαμε την εμπειρία όλων αυτής, αυτού του ρυθμού μετανάστευσης μόνο στις αρχές του δεκαετίας του 60-70 του περασμένου αιώνα. Γι' αυτό ακριβώς και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι συστάσεις αναχώρα να αντικατοπτρίζουν αυτήν την ανάγκη ευελιξίας ε, και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των διαφόρων μηχανισμών που υπάρχουν που προωθούν την ανάκαμψη και την απασχόληση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Πορτογαλίας αυτό το θέμα τονίζεται ακόμη περισσότερο εφόσον το πρόγραμμα σταθερότητας που παρουσιάστηκε από την Πορτογαλική κυβέρνηση φέτος τον Απρίλιο έχει συσταθεί από μια κυβέρνηση που είναι στο τέλος της θητείας της. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τηρεί, ε, μάλλον αναφέρεται στην περίοδο μέχρι το τέλος του 2019 σύμφωνα με τους ε, θεσπισμένους κανόνες, αλλά ε, στην ουσία η κυβέρνηση είναι στο τέλος της θητεία της γιατί σε δύο εβδομάδες μέσα στο πλαίσιο της πλήρωσης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών μας θα πρέπει να κρίνουμε αν αυτός είναι ο καταλληλότερος δρόμος ή όχι. Και γι' αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα πρέπει να προσαρμοστεί όπως για την Πορτογαλία ή με τους γείτονες της Πολωνίας που θα έχουμε, ε, θα έχουμε εκλογές τον επόμενο Οκτώβριο, θα πρέπει να προσαρμοστεί λοιπόν το ε, μερολόγιο υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο, αντικατοπτρίζοντας ενδεχομένως τις αλλαγές ε, των πολιτικών επιλογών στη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, να προσαρμοστεί με το εθνικό πρόγραμμα και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αυτό είναι μια βεβαιότητα. 15 Οκτωβρίου δεν υπά, θα υπάρχει προπολογισμό, γιατί δεν θα ε, είναι δυνατόν να ολοκληρώσετε η διαδικασία. Άρα, πώς αυτό το πλαίσιο θεωρούμε πως είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτήν την διαδικασία μέσα στο πλαίσιο μιας Ευρώπης που αντιστοιχεί στους ιδρυτικούς της στόχους, δηλαδή ανάπτυξη και αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρον. Πώς θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα τη 15 η Οκτωβρίου. Γιατί είναι, έχει προθεσμία σύμφωνα με την νέα νομοθεσία. Υπάρχουν συγκεκριμένα διαδικαστικά βήματα που σχετίζονται στενά με αυτές τις προθεσμίες. Δεν ξέρω πώς θα αυτό το πρόβλημα στη χώρα σας. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να το λύσετε. Τι θα γίνει. Uh, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε. Κοιτάξτε, οι εκλογέ είναι στι 4 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου δεν θα έχουμε προλάβει καν να συστήσουμε τη νέα κυβέρνηση. Και σίγουρα δεν θα υπάρχει νέο προπολογισμό. Και θα πρέπει, δεν είναι μόνο πρόβλημα τη Πορτογαλία και για την Πολωνία ισχύει αυτό. Γιατί και η Πολωνία έχει εκλογέ στα τέλη Οκτωβρίου νομίζω. Θα πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνε του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την πολιτική τον πολιτικό προγραμματισμό της κάθε χώρας. Καλύτερα είναι λοιπόν να ρωτήσουμε την Κομισιόν γιατί πώς θα μπορέσει να προσαρμόσει το εξάμεινο στις εκλογές μας. Ευχαριστώ. Ο Πιέρα Λεκηγέ από την Γαλλική Εθνοβουλή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας πω βεβαίως ότι χαίρομαι που διεξάγονται αυτές οι συνεδριάσεις. Με, εμείς στην Εθνοβουλή μαζί με το Γερουσία αποφασίσαμε να κάνουμε συνεδριάσεις με τους ευρωβουλευτές μας ώστε να υπάρχει συνεργασία. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά θετικό αυτό ο διάλογο. Θα ήθελα μάλιστα να εγκρίνω τι προτάσει τη έκθεση, ιδιαίτερα όσον αφορά το γεγονό ότι θα πρέπει να έχουμε τα έγγραφα τρει μήνε πριν Διότι αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στα εθνικά κοινοβούλια, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε τα κείμενα και να έχουμε τις παρατηρήσεις μας πριν από τις συστάσεις της Κομισιόν. Μάλιστα να τονίσω ότι είμαι εγώ στην αντιπολίτευση. Ίσως αυτό να φανεί και από τα όσα θα πω, Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι από την εμπειρία μου Καταρχήν διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς, αλλά αυτό ισχύει γενικότερα, γιατί το είπατε και εσείς πριν από λίγο, ότι περίπου 12% από τις συστάσεις μόνο ακολουθούνται στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι στη Γαλλία αυτό το ποσοστό είναι ακόμη χαμηλότερο. Εάν δει κανεί τον κατάλογο των συστάσεων που έχουν ε, σταλεί προς την Γαλλία, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανένας τομέας ε, στον οποίο να έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος. Για να παραθέσω τα όσα λέει ο πίνακα. Θέλω να επιμείνω λοιπόν στο γεγονό ότι είναι απαραίτητο οι συστάσει αυτέ να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη. Έχετε δίκιο όταν λέτε και νομίζω ότι είναι το σημείο υπαριθμών 16 της έκθεσης ότι όλα αυτά εξαρτώνται επίσης και ίσως κυρίως από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ωστόσο θα σας δώσω το παράδειγμα της δικής μας Βουλής για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, δηλαδή τις προθέσεις από οικονομική και δημοσιονομική άποψη όπως και η. Ε, προβλέψεις για μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ψηφοφορίας για μας. Ίσως να είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι αλήθεια. Μάλλον επειδή η πλειοψηφία φοβόταν ότι δεν θα κατάφερνε να τα υπερψηφίσουμε. Ωστόσο, είναι και μεγά... πολλή δουλειά. Και εμείς ε, στην Βουλή μας δεν μπορέσαμε να ψηφίσουμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο παρά τις διαμαρτυρίες μας βέβαια. Να επιμείνω επίσης για το γεγονός ότι είναι μεγάλη συζήτηση οι συστάσεις όταν για παράδειγμα λένε μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού καθεστώτος, μεταρρύθμιση του δικαιώματος στην εργασία έχουμε δύο είδων αντιδράσεις. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι ναι πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρουμε και υπάρχουν και από την άλλη πλευρά εκείνοι που λένε μα τι θα πει τι είναι αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έρχεται να αναμειχθεί στις δικές μας εθνικές υποθέσεις. Από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη λογική, προφανώς και δεν θα σημειωθεί πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ θα ήμουν υπέρ ο διάλογος να είναι πολύ πιο καρποφόρος και να καταλήγει σε αποφάσεις οι οποίες να είναι σύμμορφες προς την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη. Το συμφωνούσα μάλιστα να πάμε προς μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Μάλιστα μου φάνηκε μυστήριο που ακούστηκαν επικρίσεις αποκλειστικά έναντι όσων έχουν την καλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Πριν από λίγο άκουσα επικρίσεις προς τη, έναντι της Γερμανίας. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη ανταγωνιστικότητα και κοινωνική και δημοσιονομική σύγκληση. Χρειάζεται μια κοινή βιομηχανική πολιτική. Και όλα αυτά συμφωνούμε όλοι εδώ νομίζω. Χρειάζεται να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ενώ όταν βλέπουμε συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο δεν ακολουθούν οι συστάσεις της Κομισιόν και δεύτερον τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα στα εθνικά τους κοινοβούλια, θα πρέπει να ανησυχούμε για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσπάθεια ανταγωνιστικότητας και σύγκλησης. Διακόπτει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Ναι, ξέρω, ε, τελειώνω, τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε ε, και πάλι στο Ευρωκοινοβούλιο ο κύριος Τόλογιαν. Έλκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως βλέπουμε πως το ευρωπαϊκό εξάμεινο γίνεται ένα αποτελεσματικό μέσο συντονισμού οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Θα ήθελα όμως εδώ πέρα να την προσοχή σας σε ένα ασθενές σημείο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γύρω στην Άνοιξη οι κυβερνήσεις πρέπει να στείλουν στην Κομισιόν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα προγράμματα σύγκλησης ή σταθερότητας. Μετά, όπως ξέρετε, ακολουθεί η σύσταση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, σε αρκετά κρατημέλη οι εθνικές ε, κυβερνήσεις ε, δεν ε, συμβουλεύονται τα εθνικά κοινοβούλια για τα προγράμματα αυτά. Και αυτό το πρόβλημα είναι πρόβλημα δημοκρατίας, δοσίας των κυβερνήσεων στα κοινοβούλια. Τι συμβαίνει λοιπόν μετά. Τα εθνικά κοινοβούλια μαθαίνουν τα προβλήματα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις ή τη σύγκληση ή τα προγράμματα σταθερότητας ή τις συστάσεις του Συμβουλίου τα μαθαίνουν αυτά μόνο το φθινόπορο όταν οι εθνικές κυβερνήσεις παρουσιάζουν σχέδια προϋπολογισμού και συνήθως κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχεδίων προϋπολογισμού δεν υπάρχει περιθώριο να αλλάξουν τα πράγματα οπότε θεωρώ ότι για να ενισχυθεί η δημοκρατία και η λογοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων στα κοινοβουλία πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να εμπλακούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο από την άνοιξη ήδη, από την αρχή, όταν καταρτίζονται αυτά τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ Μαρία Ζωάο Ροντρίκες από τους Σοσιαλδημοκράτες. Πρέπει να πω πως συμφωνώ πλήρως με την τελευταία παρατήρηση. Είναι σημαντικό οι εθνικοί βουλευτές να εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή νωρίτερα. Όταν η Κομισιόν δηλαδή βγάζει τις εκθέσεις ε, αναχώρα και αρχίζει η κυβέρνηση να καταρτίζει τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Θέλω να σου πω εγώ την άποψή μου ως Ευρωβουλευτής. Οι συστάσεις αναχώρα στόχο έχουν τη μείωση των ανισορροπιών και οπωσδήποτε γνωρίζουμε πως αυτό απαιτεί εθνικές προσπάθειες επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αλλά βλέπουμε επίσης και τα τελευταία χρόνια ε, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα πως εάν θέλει κανείς να μειώσει τις ανισορροπίες πρέπει να ισορροπήσει και το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και συγκεκριμένα όταν μιλάμε για την Ευρωζώνη. Γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να αναπτύξουμε και έναν διάλογο μεταξύ Ευρωπαίων και Εθνικών Βουλευτών ε, επί του θέματος της έκθεσης ε, της λεγόμενης των πέντε προέδρων που κάνει προτάσεις ακριβώς για το πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί και να εξισορροπήσει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αν δούμε το παράδειγμα των επενδύσεων, ναι, Άρα έχουμε επενδύσεις ως βασική προτεραιότητα στο μείγμα πολιτικής μας. Μπορούμε όμως πως, να πούμε πως όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, ίσους όρους όσον αφορά τις επενδύσεις. Όχι. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να εξοπλίσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση με τα μέσα εκείνα που λείπουν ακόμα για να μπορούν όλες οι χώρες της ε, Ευρωζώνης να ε, προσελκύσουν επενδύσεις στο ίδιο επίπεδο. Βεβαίω τώρα έχουμε ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο, αλλά θεωρώ πως αργά ή γρήγορα, ακριβώς επειδή θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή δημοσιονομική πειθαρχία και αντιλαμβανόμαστε τα όρια των εθνικών προϋπολογισμών, αργά ή γρήγορα πρέπει να υπάρξει μια κοινή δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωζώνη. Δεύτερο παράδειγμα είναι η ανάγκη να στηριχτεί η ζήτηση μέσω του κατάλληλου μείγματος πολιτικής. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει μια οργανωμένη συζήτηση για την κατάλληλη δημοσιονομική στάση της Ευρωζώνης. Ε, ένα άλλο παράδειγμα. Η ανάγκη εμβάθυνσης του διαλόγου μεταξύ εθνικών και ευρωπαίων βουλευτών και εδώ φαίνεται. Και τέλος πρέπει να προλάβουμε τον κίνδυνο να έχουμε έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω όταν μιλάμε για ε, τα κοινωνικά. Εντάξει, προσπαθούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, είναι προς το κοινό μας συμφέρον, αλλά πρέπει να φροντίσουμε η ανταγωνιστικότητα να επενδύσεις στην ψηφιακή επανάσταση αντί να μειώνει τις κοινωνικές προδιαγραφές. Και εδώ πέρα ακριβώς πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Πώς μπορούμε δηλαδή να διασφαλίσουμε πως η κοινή μας προσπάθεια για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα δεν θα μεταφραστεί σε ε, μια μείωση της κοινωνικής προστασίας. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα για τον επόμενο διάλογο που θα είναι αρκετά εντατικός να δούμε το θέμα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Κλάους Μπάρτελ από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Γερμανία υπάρχει ευρύτατη συνέντευξη για την αναγκαιότητα του δημοσιονομικού συντονισμού, αλλά πρέπει να δούμε ψύχρεμα τα αποτελέσματα και να δούμε το εάν ε, πηγαίνουν προς τα εκεί που θέλουμε. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως πέρα από την έλλειψη ανάπτυξης αυξάνονται οι ανισότητες μεταξύ κρατών μελών αλλά και εντός των κρατών μελών μεταξύ περιφερειών και κοινωνικών τάξεων. Γι' αυτό θεωρώ πως θα ήθελα να αφαιρθώ λίγο στο παράδειγμα της ε, Γερμανίας και των συγκεκριμένων συστάσεων. Αν είχαμε ακολουθήσει τις συστάσεις αυτές το 2008 δεν θα είχαμε ξεπεράσει την κρίση όπως το κάναμε. Εμείς κάναμε το αντίθετο από τις συστάσεις. Σταθεροποιήσαμε και δεν απορριθμίσαμε την αγορά εργασίας. Ενισχύσαμε τους κοινωνικούς εταίρους και αυξήθηκε η εσωτερική ζήτηση κατά 2% του ΑΕΠ και έτσι προωθήθηκε και η ανάπτυξη και δεν ε, ελαστικοποιήσαμε την αγορά εργασίας όπως προτείνονταν. Και αν ξαναδούμε τις συστάσεις που έγιναν στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, σε αντίθεση με την συζήτηση για τα πλεονάσματά μας, διαπιστώνω πως η ίδια φιλοσοφία η νεοφιλελεύθερη χρησιμοποιείται για τη Γερμανία όπως και για ασθενέστερες χώρες και πραγματικά απορώ για το ότι κατηγορεί κανείς ε, τη Γερμανία για το ότι δεν τηρεί το φρένο χρέους, ότι οι υπηρεσίες λέτε δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές και επιπλέον ζητάτε να αυξηθεί η κατανάλωση και να, με συγχωρείτε να φορολογηθεί περαιτέρω η κατανάλωση. Μα αν γίνει αυτό θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πλεόνασμα. Εμείς θα περιμέναμε έναν έπαινο για το ότι εισήχθη βασικός μισθός και ενισχύσαμε τα συνδικάτα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για το ότι οι επενδύσεις και το συνταξιδοτικό σύστημα ενισχύθηκαν. Δεν θέλουμε να μειώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε την ισορροπία για να ενισχύσουμε εισαγωγές και την κατανάλωση. Οι συστάσεις όμως πήγαιναν στην αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε πως έχουμε μια ιδεολογική κατεύθυνση και δεν κοιτάει κανείς τη συγκεκριμένη κατάσταση. Επίσης θεωρούμε και οπωσδήποτε και αυτό είναι και αντικείμενο της εσωτερικής πολιτικής συζήτησης πως οι συστάσεις πρέπει να έχουν διαφορετική κατεύθυνση αν θέλουμε επενδύσεις στην Ευρώπη και δεν πρέπει να αφήσουμε να αυξηθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Πρέπει να δούμε και την δυνατότητα του κράτους να δράσει ε, στον τομέα της οικονομίας. Δεδομένης λοιπόν της ε, ασφαλούς κατάστασης ε, στην παγκόσμια οικονομία πρέπει να ενισχύσουμε την εσωτερική μας οικονομία να επενδύσουμε και να τονώσουμε την εσωτερική ζήτηση στην Ευρώπη. αντί να εξάγουμε συνεχώς. Τρίτον, να διαβάσουμε τις συστάσεις. Πρέπει να μειωθεί η φορολογία της εργασίας και να μην φορολογούμε τους καταναλωτές αλλά να πάμε σε μια κοινή φορολογία του κεφαλαίου και έναν φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Τέταρτον, δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για ελαστικότητα, αλλά κυρίως για ασφάλεια και για όρους και ερισιμότητα. Και τέλος για τη συζήτηση ε, στη, της μετανάστευσης και την τρέχουσα κατάσταση. Βλέπουμε, σε αυτής της ε, κατάστασης, θα πρέπει να ρυθμίσουμε περισσότερο την κατάσταση στην αγορά εργασίας γιατί η μετανάστευση και η περαιτέρω αταξία θα έλεγα στα κοινωνικά συστήματα δεν ε, πάνε μαζί. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ε, για τα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα σχόλια, σχόλια σας. Ο κύριος Κριστόφ Ματσνέτερ από την Αυστρία παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συνάδελφο. Άκουσα και τον κύριο Χίρτε. Ε, όταν ασκούμε κριτική στο εμπορικό ισοζύγιο, δεν σημαίνει ότι ασκούμε κριτική στις εξαγωγές αλλά στο ότι δεν υπάρχει αρκετή αγοραστική δύναμη στο εσωτερικό της οικονομίας. Και το οποίο βεβαίω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω και τα ελλείμματα. Τώρα, για το Sixpack θεωρώ πω η κατάσταση είναι ξεκάθαρη η Ευρώπη στη διεθνή ανταγωνισμό δεν τα πάει καλά και αυτό ακριβώς ε, το κομμάτι αν δούμε τις υπόλοιπες περιοχές ε, του κόσμου είναι εκεί που δεν τα πάμε καλά και εδώ πέρα πρέπει να ρωτηθούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε Οπότε υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσει, αλλά δεν αναρωτιόμαστε γιατί από την πλευρά των εσόδων δεν έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, να φορολογήσουμε δηλαδή τα κέρδη τα οποία δημιουργούνται εδώ πέρα, να τα φορολογήσουμε εδώ πέρα. Ας δούμε τη φορολογία την εταιρική στις ΕΠΑ ή στην Κίνα με την ευρωπαϊκή. Πόρο απέχουν. Και αν δούμε και τα LuxLeaks, Πραγματικά βλέπουμε τεράστια έλλειψη. Δεν καταφέραμε δηλαδή να μετατρέψουμε την ευρωπαϊκή δημιουργία αξίας σε φορολογικά έσοδα. Όσον αφορά το ζήτημα της απορρίθμισης, π.χ. το ότι δεν εφαρμόζονται, δεν υπάρχει αρκετή άρση των εμποδίων στην άσκηση των επαγγελμάτων. Μα πρόκειται για πράγματα τα οποία ισχύουν εδώ και αιώνες, να μην πω και μια χιλιετία και είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτό το οποίο λέμε ευρωπαϊκή ποιότητα και όσον αφορά τη Γερμανία και τη χώρα μου την Αυστρία και ακριβώς αυτή η ποιότητα ε, οδηγεί την ε, βιομηχανία να είναι ανταγωνιστική με υψηλές τιμές με την απορρίθμιση θα καταργηθούν ορισμένα επαγγέλματα και ελπίζουμε μετά ότι κάτι θα βρει αγορά να τα αντικαταστήσουν. Μα τι θα γίνει στο τέλος, κανείς δεν θα εκπαιδεύει νέες γενιές ε, να αναλάβουν την ε, δουλειά του. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε ένα σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε όπως είπα σε βάθος αιώνων το οποίο σημαίνει πως θα πρέπει κανείς να φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας πριν μπορέσει να βγει στην αγορά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ίσως να είναι δικαιολογημένη η αντίσταση κάποιων ε, κρατών μελών. Να δοθούν έτσι δηλαδή κίντρα στους νέους να μάθουν ένα επάγγελμα για να βρουν μετά μια δουλειά. Βεβαίως, Μιλάμε και για κάποιες ε, ηθικές απαιτήσεις ε, τις οποίες ε, έχουμε όταν μιλάμε για την εξάσκηση ενός επαγγέλματος. Εγώ προσωπικά ας πούμε είμαι φοροτεχνικός και σύμβουλος ε, επιχειρήσεων. Και εμείς δεν έχουμε καταφέρει εδώ πέρα βεβαίως ε, να φτάσουμε παραδείγματος χάρη τις ε, τέσσερις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες με δικές μας εταιρείες. Λοιπόν, η δικιά μου η έκκληση στους συναδέλφους του ΕΛΚ είναι ασκήστε πίεση περισσότερη πίεση. Συζητάμε 20 χρόνια για μια εσωτερική αγορά εντός της νομισματικής ένωσης. Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται και μια κοινή φορολογική ε, βάση και δεν είναι δυνατόν να φορολογούμε μόνο την εργασία. Πέντε λεπτά ακριβώς σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να εργαστεί πολύ σκληρά για θέματα ε, φορολόγησης και να εργαστεί έτσι ώστε να προχωρήσουν τα ε, μέτρα CCCTB και ασκεί πίεση για αυτό. Φορ Νέπαρ τώρα από την Ουγγαρία. Για την κοινή φορολογική εταιρική βάση δηλαδή. Ο εκπρόσωπος της Ουγγαρίας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εκ μέρους του Ουγγρικού Κοινοβουλίου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δώσατε σε μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων να πάρουν το λόγο και να σχολιάσουν για την οικονομική πολιτική και τα προγράμματα που ε, υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν μετά την, το ξέσπασμα της κρίσης το 2008. Με βάση την εμπειρία μας τα περασμένα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει βελτιώσει τα μάλα την κατάσταση δίνοντας πολλές ευκαιρίες στα κράτη-μέλη να σχολιάσουν αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, οφείλουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να αυξήσουμε τις ευθύνες των εθνικών κοινοβουλίων στο σκέλος της εφαρμογής. Όσον αφορά τις ειδικέ συστάσεις ανά χώρα, θα πρέπει αυτές να επικεντρώνονται σε ζητήματα πολιτικής. Σε γενικές γραμμές καλωσορίζουμε την ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι μια εξέλιξη ε, την οποία θεωρούμε ευπρόσδεκτη και ε, θέλουμε και καλωσορίζουμε την πιο εστιασμένη και συγκεκριμένη διατύπωση των συστάσεων αναχώρα. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ευρύ περιθώριο στα εθνικά κοινοβούλια και αναφέρεται αυτό στο προήμιο. Θα πρέπει και το προήμιο και οι αιτιολογικές σκέψεις να διευκρινιστούν. Η υποβολή γραπτών σχολείων θα πρέπει να επιτρέπεται και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε διαβουλεύσεις. Η Ουγγαρία καλωσορίζει τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το έλλειμμα του προϋπολογισμού παραμένει κάτω από το 2,5% και στο 2016 και συμφωνούμε επίσης στο ότι οι στόχοι των εθνικών προγραμμάτων θα πρέπει να είναι καλύτερα εστιασμένοι. Ωστόσο, πρέπει να δούμε πώς θα αναδιαμορφωθεί το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να εκπληρώσει τους στόχους του πραγματικά και να έχει περισσότερη προστιθέμενη αξία. Τα ζητήματα που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ήταν ανέκαθεν στην ε, ε, μερίσια διάταξη του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Τα εξετάζουμε στενά. Αρχής γενομένης από το 2012 έχουν δημοσιευθεί εκθέσεις και η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα σύγκλησης το οποίο στείλαμε στα αρμόδια και αντίστοιχα όργανα και είχαμε και ακροάσεις μετά τις ειδικέ ε, συστάσεις αναχώρα. Ως προς τις συστάσεις του 2015, το Μάιο έγινε μία διαβούλευση στη Βουδαπέστη με την κυρία Γελασκόβα, η οποία είναι υπεύθυνη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Η Άννα Μπίρχαλα από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σε αυτό ε, ε, την πολύ σημαντική, συζήτηση και θα ήθελα να μιλήσω στα ρουμανικά. Αναλύουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και κυρίως τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ε, το ότι η νέα Προεδρία αντιμετωπίζει με ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει με πολύ ανοιχτό τρόπο και ευρύ ε, με διευρυμένους ορίζοντες τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ενθαρρυνεί και να εμβαθύνει το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και καλωσορίζουμε και τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι έχει να κάνει με την απλούστευση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δίδεται έμφαση σε μικρό αριθμό προκλήσεων και προτεραιοτήτων και δημοσιεύεται η ανάλυση για κάθε χώρα τρεις μήνες νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και έτσι μπορούμε να αναλύσουμε τα πράγματα έγκαιρα και σε βάθος εμείς στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας και τα μέλη αυτής της Επιτροπής παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αρχής γενομένης της έκθεσης για την ανάπτυξη και ε, των ε, συστάσεων αναχώρα. Εκδίδουμε γνωμοδότηση και αναγνωρίζουμε ότι πράγματι είναι ανάγκη να ενισχύσουμε την συσσωρευμένη αθρηστική ζήτηση και όχι μόνο την ε, συσσωρευμένη αθρηστική προσφορά. Η συνιστόσα της ανάπτυξης είναι ε, πολύ σημαντική και θα πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις, ε, δημοσιονομική πειθαρχία και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο Juncker και η προσέλκυση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι κάτι το καλό. Το έχουμε συζητήσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή στη Ρουμανία και έχουμε προτείνει να γίνει και ένας δημόσιος διάλογος μετά από την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέπουν να εκπληρώσουμε τους οικονομικούς και κοινωνικούς μας στόχους. Θα πρέπει αυτούς τους στόχους να τους ακολουθήσουμε σε εθνικό επίπεδο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Προτεραιότητα είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Στη Ρουμανία έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το νέο φορολογικό κώδικα που ε, θα πρέπει ε, να εξεταστεί. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σωστή μεταξύ της φόρο ε, απαλλαγής από τη μία, της φορολογικής ελάφρυνσης μάλλον και της ανέπτυξης από την άλλη. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε προς την φορολογική ελάφρυνση και να φτάσουμε το έλλειμμα του 1,5% το 14. Ε, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι σημαντική στην Ρουμανία και πρέπει να εξετάσουμε τις ειδικές ανάγκες μιας οικονομίας η οποία ε, ε, αποκλίνει αρκετά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο νέος φορολογικός και δημοσιονομικός κώδικας μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε τα νέα μέτρα για φόρο απαλλαγές. Έτσι θα αξιολογήσουμε την οικονομική συμπεριφορά και έτσι μπορούμε να ενθαρρύνουμε και την προσφορά και την ζήτηση. Αυτά συνοδεύονται από διαρθρωτικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί το ΑΕΠ. Οι οικονομικές επιλογές θα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο και να εμπλέκονται τα εθνικά κοινοβούλια. Θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εμπλέκονται σε αυτή τη διαβούλευση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνάντηση η οποία είναι απόδειξη διαφάνειας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Πρόεδρος, η κυρία Λέτς από τη Γερμανική Βουλή. Ευχαριστώ και Ζήνη Λέτς, είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και μέλος των ε, αριστερών. Μίλησαν ήδη δύο συναδελφοί μου, τόνισαν διαφορετικά πράγματα, αλλά ανήκουν και οι δύο στον κυβερνητικό συνασπισμό. Εγώ είμαι της αντιπολίτευσης. Στη Γερμανική Βουλή συζητάμε ήδη τον ε, προϋπολογισμό. 312 δισεκατομμύρια ευρώ είναι και υποθέτω πως θα πρέπει να αυξηθεί. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί οι κανόνες και οι συστάσεις ε, θα πρέπει να προσαρμόζονται και στις προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε. Το ανέφερε ο κύριος Μπάρτελ, θέλω να το πω και εγώ. Εγώ είμαι πεπισμένη πως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πώς θα απαντήσουμε στην πρόκληση των προσφύγων πολέμου που κατευθύνονται στη Γερμανία τη Σουηδία και τις άλλες ε, χώρες. Και οπωσδήποτε η κατάσταση αυτή θα έχει επιπτώσεις ε, και στην ε, πολιτική, την οικονομική, του προϋπολογισμού και τις φορολογίες. Και βεβαίω θεωρώ πως τα κάτι μέλη θα πρέπει να θέσουν το ερώτημα τι μπορούν να κάνουν για να σταματήσουν οι αιτίες που δημιουργούν πρόσφυγες και άρα είμαι πεπισμένη πως όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και η Γερμανία πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσουν τις εξαγωγές όπλων σε περιοχές κρίσης. Βεβαίως, έχουμε το θέμα των επενδύσεων. Αν έχω καταλάβει καλά τη συζήτηση, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να ε, γίνουν επενδύσεις. Το θέμα είναι βεβαίως τι εννοεί ο καθένας εδώ πέρα όταν μιλάμε για σημαντικές επενδύσεις ποια είναι μια μεγάλη επένδυση και ποια είναι μια μικρή επένδυση ο κύριος Μπάρτελ σωστά υπενθύμησε πως στη Γερμανία το 2008 εμείς ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην Γερμανία και τώρα πράγματι έχουμε άλλο ένα πρόγραμμα το οποίο έχει στόχο να προλάβει διάφορες εντάσεις. Βεβαίω, το άλλο θέμα είναι το θέμα του χρέους. Θεωρώ πως ε, στη Γερμανία συμφωνούμε πως δεν πρέπει να γίνονται χρέη, να αναλαμβάνονται χρέη που δεν χρειάζονται. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα πως σημαντικό κομμάτι της αποφυγής δημιουργίας χρέους είναι ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα και να φορολογεί κανείς ε, πρώτα απ' όλα κλείνοντας τα παραθυράκια αλλά βεβαίως και να διαμορφώσει το σύστημα έτσι και βεβαίως και να εξηγιάνει του προπολογισμούς. Τέλος, όσον αφορά αυτά τα οποία είπε ο βουλευτής ο κ. Ντιμάζο για την ε, έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Γερμανικής Βουλής ε, για το θεσμικό πλαίσιο του Eurogroup και για το αν έχει καν το δικαίωμα να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις με κάποια μόνο και όχι όλα τα μέλη. Και θεωρώ πως ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας απασχολήσει και στο Κοινοβούλιο και στο Eurogroup. Έχουμε πολλά επίσημα φόρα, έχουμε συνθήκες και την νομιμοποίηση μέσω κανόνων, αλλά άλλα φόρα δεν έχουν αυτή την νομιμοποίηση και πρέπει να υπάρξει κάποια διόρθωση. Και τέλος, ένα αστιάκι, αν μου επιτρέπετε. παρουσιάστηκε αυτή η έκθεση της ε, γερμανικής, ε, της επιστημονικής υπηρεσίας της ε, Βουλής και βλέπω πως ε, παρουσιάστηκε παντού στον τύπο. Την εκτιμούν από ό,τι φαίνεται περισσότερο και από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ. Ο Γάλλος γερουσιαστής ο κύριος Ντέμον Γκολφιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ο συνάδελφος που μίλησε προηγουμένως και εγώ είμαι μέλος της αντιπολίτευσης και θέλω να πω ότι η Γαλλία είναι μία από τις δύο χώρες που ε, αυξήθηκε το έλλειμμα τα τελευταία χρόνια και οι άλλες χώρες είχαν τα, τις δημόσιες δαπάνες να αυξάνονται κατά 1,2% το χρόνο, ενώ στη Γαλλία αυτές αυξάνονταν κατά 2,5% το χρόνο, διπλάσια αύξηση δηλαδή. Ο δυστυχώς το πρόγραμμα σταθερότητας που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο δεν τηρεί ε, τις ε, δεσμεύσεις δημοσιονομικής προσαρμογής που εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι διαφορετική η προσέγγιση ε, της γαλλικής κυβέρνησης από τη μία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την άλλη. Οι υποθέσεις εργασίας δεν είναι ίδιες που ε, υιοθετούν οι δύο αυτοί φορείς. Άρα η ερώτησή μου είναι απλή. Πώς θα διασφαλίσουμε στο μέλλον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν κοινή βάση υπολογισμού και άρα τελικά ε, θα ε, τηρηθούν τα δέοντα. Για παράδειγμα, ως προς το ε, διαρθρωτικό έλλειμμα, η Γαλλία το υπολογίζει διαφορετικά από ό,τι το υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι μιλούμε την ίδια γλώσσα. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο πολλοί άλλωστε το έχουν αναφέρει, πώς θα εμπλακούν περισσότερο και καλύτερα τα εθνικά κοινοβούλια, όχι μόνο στην ε, ε, παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της σταθερότητας, αλλά πώς θα εμπλακούν στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής. Από πιο νωρίς, από πιο προκαταρκτικό στάδιο. Σίγουρα είναι χρήσιμε τέτοιου είδου συναντήσεις όπως η σημερινή. Καλό θα ήταν όμως να έχουμε και διμερείς συναντήσεις μεταξύ ε, κοινοβουλευτικών ε, επιτροπών διαφόρων εθνικών κοινοβουλίων. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Οικονομικών της Γαλλική Γερουσίας θα είχε ενδιαφέρον να συναντηθεί με κάποιου ομολόγου τη από το Πορτογαλικό Ισπανικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα. Ε, Όλα αυτά θα ήταν χρήσιμα, είναι ε, εκείνη τα πραγματικά ερωτήματα και οι συνεδριάσεις σαν τη σημερινή μας βοηθούν ιδιαίτερως. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, να δώσω το λόγο στον κύριο Μαριά από την Ελλάδα. Πέντε λεπτά έχετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πολύ σημαντική η συνάντηση που έχουμε με τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια διότι πιστεύω ότι έτσι διαμορφώνουμε ένα διάλογο και μπορούμε σιγά σιγά να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα. Διότι τόσο τα Εθνικά Κοινοβούλια όσο και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκφράζουν τους λαούς της Ευρώπης. Και επομένως νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά σε σχέση με την ε, Ευρώπη των τραπεζών, η οποία πλέον είναι αυτή που κυριαρχεί επί των πολιτικών των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πολλά κοινά απέναντι στην ίδια την Επιτροπή, την Κομισιόν, η οποία και αυτή ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που ονομάζουμε γραφειοκρατία των Βρυξελών. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντική τη συνάντηση αυτή γιατί μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις και κυρίως γιατί μπορούμε να γνωριστούμε στην πράξη. Διότι αν δεν υπάρχει και αυτή η, γνώση του ενός απέναντι στον άλλο, νομίζω ότι δεν έχουμε μια σαφέστατη εικόνα για το τι μιλάμε και ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε. Δεύτερο, αυτό που άκουσα από τον συνάδελφο από τη Γαλλία, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και των εθνικών κοινοβουλίων, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ μέχρι πέρυσι ήμουν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ξέρετε στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και του α, πρωτοκόλου για την επικουρικότητα τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συνεργάζονται και μάλιστα να βάζουν και βέτο εάν διαμορφώσουν ένα αριθμό εθνικών κοινοβουλίων, μία πορτοκαλί κάρτα όπως λέγεται, απέναντι σε νομοθετικές πρωτοβουλίες της ίδιας της Κομισιόν. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ σημαντικό και το να υπάρχει και η άμεση συνεργασία των ίδιων των εθνικών κοινοβουλίων. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο ποιε είναι οι αρμοδιότητε. Διότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο αφορά την άσκηση οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική ανήκει στι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η νομισματική πολιτική. Επομένω, πρόκειται για μια διαδικασία συντονισμού και συνεργασίας αλλά τον τελευταίο λόγο το, στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου την έχουν τα κράτη-μέλη και την έχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ιδίω δε για του προπολογισμού δεν μπορεί να νοηθεί η δημοκρατία χωρί τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν την αρμοδιότητα να καθορίζουν κυρίαρχα τον προπολογισμό του. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο με στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και αυτά που σα λέω τα έχω πει και σε προηγούμενη συνεδρία εδώ στην Επιτροπή ε, Οικονομική και Νομισματική Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι παρατηρώ ότι εκ μέρου τη Κομισιόν υπάρχει μια προσπάθεια υφαρπαγή αρμοδιοτήτων που εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να ανήκουν στα κράτη-μέλη. Αυτό σε σχέση με το ρόλο και το πώ πρέπει να συνεργαζόμαστε. Έθελα επίσης να επισημάνω ότι στις χώρες οι οποίες βρέθηκαν σε μνημόνιο σε μεγάλο βαθμό έχει ανατραπεί και η ίδια διαδικασία λειτουργίας των Εθνικών Κοινοβουλίων. Διότι οι αποφάσεις παίρνονται στην ουσία από την Τρόικα, η οποία εάν δεν εφαρμόσει ένα κράτος μέλος το οποίο βρίσκεται σε μνημόνιο, σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, αυτό που επιβάλλει η Τρόικα, πολύ απλά σταματάει τη χρηματοδότηση, σταματάει το να δίνει δάνεια Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων επιβάλλει την πολιτική της η Τρόικα σε κυρίαρχα κράτη και φυσικά ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων γίνεται δευτερεύον. Και αυτό το βλέπουμε και στις αποφάσεις του Eurogroup, το οποίο δεν είναι εκλεγμένο όργανο, στην ουσία είναι ένα άτυπο όργανο, το οποίο όμως παίρνει κυρίαρχες αποφάσεις. Και αν έρθετε στην περίπτωση της Ελλάδας που είναι καταξοχήν περίπτωση όπου το Eurogroup έπαιρνε κυρίαρχες αποφάσεις, όπου η Τρόικα επέβαλε τις πολιτικές στην Ελλάδα και η Ελληνική Βουλή δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Όταν ήμουν βουλευτής μας έφερναν 300-400 σελίδες νομοσχέδιο και μας έλεγαν θα το ψηφίσετε σε δύο ημέρες διότι διαφορετικά δεν θα πάρει χρηματοδότηση η Ελλάδα και θα πτωχεύσει. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα εθνικό κοινοβούλιο στην τελευταία απόφαση του Ιουλίου όπου επέβαλε η Τρόικα ένα νέο μνημόνιο στην Ελλάδα, τους έστειλαν στην Ελληνική Βουλή ένα νομοσχέδιο 700 σελίδες και τους είπαν θα το ψηφίσετε σε δύο ημέρες. Κανείς δεν πρόλαβε να διαβάσει τι ψήφιζε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια παραβίαση των αρχών της δημοκρατίας με το ρόλο που λειτουργεί η Τρόικα. Και είναι θέματα σημαντικά τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Σιλβί ε, Ευχαριστώ κυρία Σιλβί Γκουλάχ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το γεγονός ότι μου δίνετε το λόγο σημαίνει ότι σας αρέσουν τα γαλλικά. Τέλος πάντων, έπαμε. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, σε ένα θέμα για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κάνει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Μετά από ορισμένα χρόνια που έχουμε πλέον εμπειρία και δώσαμε προτεραιότητα τα κατεπήγοντα μέτρα για να προασπίσουμε την οικονομική σταθερότητα, θα μπορούσαμε πλέον να προβληματιστούμε για μια καλύτερη ε, ρύθμιση σε παγκόσμιο επίπεδο του τομέα των χρηματοπιστωτικών. Θα πρέπει κανείς να δράσει σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό δημιουργεί πρόβλημα για κάθε δημοκρατία, είτε είναι οργανωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε αλλού έχουμε τον οργανισμό που ασχολούνται με τα λογιστικά πρότυπα. Έχουμε διάφορα συμβούλια και οργανισμούς σε διεθνή επίπεδα που έχουν να κάνουν με τον κόσμο των χρηματοπιστωτικών και η Ευρώπη εκπροσωπείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους σε όλα αυτά. Άρα η διαφάνεια και ο σεβασμός των κανόνων από όλους τους εταίρους δεν είναι πράγματα καθόλου σαφή. Όλα αυτά έχουν αφαιθεί στο τυχαίο. Ήθελα λοιπόν να πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή, αυτή η δουλειά και αν υπάρχουν άνθρωποι από τα εθνικά κοινοβούλια που τους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, που θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους, τις βέλτιστες πρακτικές, το πώς μπορεί κανείς να εκπροσωπηθεί καλύτερα σε όργανα τεχνικοπολιτικής φύσης. Να σας πω ότι είμαστε διατεθειμένοι και με ενθουσιασμό θα τους ακούσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις. Από εκεί και πέρα, πέρα από την εκπροσώπηση της Ευρώπης στα διεθνή όργανα και διεθνείς φορείς, θέλω να πω ότι είναι λίγο διάλογο κοφών με, με τα εθνικά κοινοβούλια δεν είναι το θέμα η δημοκρατική νομιμοποίηση η εθνική έναντι της ευρωπαϊκής νομιμοποίησης. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε στην βασική πρόκληση που είναι να ε, εμπιστευτούν ξανά οι πολίτες τους ευρωπαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς. Σέβομαι ιδιαιτέρως ορισμένες χώρες, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ορισμένες χώρες μόνο για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει λογοδοσία για όλες τις αποφάσεις στο σύνολο της ζώνης του Ευρώπου, που, αποφάσεις που επηρεάζουν θέματα εξαιρετικά κρίσιμα. Ε, χαίρομαι που ήρθατε και σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Με χαρά θα ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ντάριους Ροζάτη, παρακαλώ. Πολλά Ακούσατε και ενδιαφέροντα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ήταν ένα εξαιρετικά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συναρπαστική συζήτηση. Ευχαριστώ όλους όσοι πήραν μέρος σε αυτήν. Έχω σημειώσει όλες τις παρατηρήσεις σας, διαβεβαιώ και θα τις λάβω υπόψη μου την τελική ε, σύνταξη του κειμένου. Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε τροπολογίες και εργαζόμαστε πάνω στο τελικό έγγραφο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ή τρία ζητήματα που έχουν συζητηθεί αρκετά εντατικά και να ξεκινήσω με τη δική μου ερώτηση, την ερώτηση που έχω, δώσει εγώ στην, που έχω κάνει εγώ στην αρχή της συζήτησης, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι για αυτή την απουσία ιδιοκτησίας ε, των ειδικών ε, συστάσεων αναχώρα. Γιατί είναι τόσο χαμηλός ο βαθμός και το ποσοστό αφομοίωσης των συστάσεων αυτών. Άκουσα ε, διάφορες προτάσεις και υποδείξεις προς την κατεύθυνση αυτή και πιστεύω ότι ένα είναι σαφές σίγουρα, ότι Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία και τις διάφορες επιμέρους αλληλουχίες αυτής. Ορισμένες φωνές αναφέρθηκαν στο ότι κάποια στάδια αλληλοεπικαλύπτονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή στο γεγονός ότι ορισμένα για παράδειγμα, δεν έχουν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν και να αντιδράσουν στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, άκουσα επίσης ε, την διαπίστωση ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν ενημερώνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό πράγματι δείχνει την αδυναμία αυτού του μηχανισμού. Σε αυτή την εξάμεινη περίοδο υπάρχει αλληλεπίδραξη μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διάφορα έγγραφα πρέπει να ε, προετοιμαστούν και δεν υπάρχει ενδεχομένω χρόνος να ε, ληφθούν υπόψη. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν με αυτά και αυτό είναι μια, ένα σημαντικό συμπέρασμα που αντλώ από αυτή τη συζήτηση. Δεύτερο, είναι το εξής. Ως προς το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στη Γερμανία. Πράγματι, τα πλεονέσματα είναι καλό πράγμα. Είναι δείγμα σθένους της γερμανικής οικονομίας. Όμως έχουν ακουστεί φωνές ότι δεν είναι και τόσο επιθυμητά και τόσο ευκταία. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει συμμετρία αυτή τη στιγμή μεταξύ των ελλημάτων και των πλεονασμάτων. Καταρχάς δεν υπάρχει νομική συμμετρία. Γιατί το όριο 6% για τα πλεονέσματα είναι ενδεικτικό, ενώ το έλλειμμα, το όριο του 3% είναι νόμος. Είναι νόμιμο όριο. Άρα δεν υπάρχει συμμετρία, δεν υπάρχει κάτι το αντίστοιχο. Και πρέπει αυτό να το πούμε. Μια χώρα που έχει έλλειμμα είναι σε πολύ υψηλότερο κίνδυνο να βιώσει αστάθεια εάν υπάρξει ε, διακοπή του κεφαλαίου, της ροής αυτού ε, που χρηματοδοτεί αυτό το έλλειμμα. Και βεβαίως αυτό δεν είναι τόσο πρόβλημα για την πλεονισματική χώρα η οποία είναι σε πολύ πιο ασφαλή θέση. Ωστόσο, μιλώντας για την νομισματική ένωση όπου οι χώρες είναι άλληλο συνδεδεμένες και δία συνδεδεμένες εξαιρετικά ε, ισχυρά και όπου μία κατάσταση μπορεί να διαχυθεί από τη μία χώρα και να επεκταθεί σε άλλη σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει έλλειμμα χωρίς αντίστοιχο πλεόνασμα και δεν υπάρχει πλεόνασμα χωρίς αντίστοιχο έλλειμμα σε κάποια άλλη χώρα. Και δεδομένου ότι το ενδοκοινωτικό εμπόριο είναι σημαντικό κομμάτι του εξωτερικού εμπορίου της Γερμανίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο πλεόνασμα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας σημαίνει αυτόματα αντίστοιχο σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών κάποιας άλλη χώρα ή κάποιων άλλων χωρών. Άρα οι χώρες, οι ελληματικέ, οι οποίες ε, καταγγέλλονται, ε, καλούνται να εξαλείψουν αυτό το έλλειμμα, αλλά αυτό είναι δύσκολο χωρί την αντίστοιχη συνεργασία από την άλλη πλευρά, από την απέναντι πλευρά. Λέω λοιπόν ότι βεβαίω ότι το ε, πλεόνασμα ενδεχομένως είναι, είναι ένδειξη ανταγωνιστικής οικονομίας, όμως εάν είσαι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε το γεγονός ότι είσαι μέλος συνεπάγεται ε, συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενδεχομένως αλλά και ε, την πιθανότητα να υποστείς διάδοση ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζονται αλλού στην ίδια ζώνη. Και όλα αυτά είναι ζητήματα προς συζήτηση. Τώρα θα ήθελα να ε, ε, βεβαιώσω τα μέλη που έχουν διαφορετική άποψη για τη λιτότητα και ενδεχομένως την κύρια και κυριαρχική άποψη ότι η έκθεση δεν, έχει, δεν αναφέρει τη λέξη λιτότητα. Είναι χιλιοπεγμένο το τραγούδι της, των παραπώνων εναντίον της λιτότητας. Καλούμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική με αντικυκλικό τρόπο για να ενθαρρύνουν τις οικονομίες τους. Μόνο βεβαίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος. Το θέμα της λιτότητας λοιπόν παρουσιάζεται με εσφαλμένη προοπτική. Κανείς ε, δεν χαίρεται με τη λιτότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως η λιτότητα ήταν πολύ απλά αναπόφευκτη, ειδικότερα στην περίπτωση των χωρών που έχασαν την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και δεν υπήρχε άλλη λύση. Δεν είναι συνταγή υπό την έννοια ότι εσείς π.χ. στην χ χώρα μπορείτε να ξοδέψετε παραπάνω αλλά εμείς σας ζητούμε να ξοδέψετε λιγότερα και άρα βεβαίως υπάρχει κίνδυνος ύφεση, κάθε περικοπή σε δημόσιε δαπάνε είναι πάγεται ύφεση. Δεν ήταν όμω αυτή η κατάσταση. Οι, οι χώρες αυτές που αναγκάστηκαν να κόψουν τι δαπάνε του, να τις περικόψουν, δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να δανειστούν από αλλού. Δηλαδή ήταν αναγκαίο. Δεν λέμε ότι είναι ένα άρετο, αλλά δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώ. Και δεν νομίζω ότι είναι πια το βασικό ζήτημα. Στην έκθεση δεν μιλούμε πια γι' αυτό. Δεν μιλούμε για την ανάγκη συνέχισης της λιτότητας. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι ότι θα πρέπει να εξηγιανθούν αυτές οι οικονομίες προστατεύοντας τις δημόσιες επενδύσεις εξ αρχής, κάταρχας. Επομένως είναι κάτι διαφορετικό αυτό που λέμε. Τώρα, ο πρόεδρος διακόπτη. Ο κύριος Ροζάτη πάλι. Αυτό ήθελα να πω. βεβαίω δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω όλες τις σημαντικές συνεισφορέ που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτή τη συζήτηση. Σημειώνω όλα αυτά που είπαν οι ομιλητές και θα προσπαθήσω να αντικατοπτρίσω τις σημαντικές τους απόψεις στο τελικό ε, προσχέδιο της έκθεσης που θα σας υποβάλω. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Πριν ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτού του σημείου του ημερήσιας διάταξη θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιε παρατηρήσεις με τη σειρά μου. Μία για την ουσία της οικονομικής πολιτικής και μία δεύτερη πιο διαδικαστική. Αυτά που είπε ο εισηγητή είναι πολύ σημαντικά. Ίσως δεν συγκλίνει η ανάλυση μας 100% για την ποιότητα της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Νομίζω όμως ότι προκύπτει συνένεση από πλευράς της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για τον σωστό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος της οικονομικής πολιτικής και της δημοσιονομικής πολιτικής για την ε, ΟΝΕ, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται μέσω αυτής της παραγράφου, για παράδειγμα, για την ε, ανάγκη αντικυκλικής πολιτικής, για την ανάγκη ε, προστασίας των, των καταθέσεων κτλ. Αλλά τώρα η Κομισιόν έχει ακολουθήσει την ουδέτερη δημοσιονομική στάση και, και κάπως μεγαλύτερη ευελιξία από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά τίνει να αντιμετωπίζει το θέμα της κοινή δημοσιονομικής στάσης της Ευρωζώνης και εδώ έχουμε και το σχέδιο Γιούγκερ για τις επενδύσεις και εδώ στο Κοινοβούλιο προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιο είναι το καταλληλότερο μείγμα πολιτικής που θα μπορούσε να εγγυηθεί γρήγορα ανάπτυξη και σταθερότητα. Αυτή η συζήτηση λοιπόν θα μπορούσε να δώσει περισσότερη όθηση στο συγκεκριμένο μακροοικονομικό στοιχείο της έκθεσης και έπειτα κάτι ακόμα το οποίο είναι πιο θεσμικό και μεθοδολογικό. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον τα σχόλια που έγιναν σε σχέση με το γεγονός ότι από τη μια πλευρά πρέπει να εξασφαλίσουμε το σεβασμό των κανόνων και την ε, επιβολή τους, ενώ απ' την άλλη πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συστάσεις είναι καλές και ότι δεν θα είναι αντιπαραγωγικές, όπως ε, ε, ανέφεραν οι Γερμανοί μας συνάδελφοι. Δεν ξέρω βεβαίω αν όλοι οι συνάδελφοι τη Bundestag συμφωνούν γι' αυτό. Πάντω το γεγονό ότι η Γερμανία είναι τώρα ανταγωνιστική συνδέεται και με το γεγονό ότι αυτή η χώρα ίσω έξυπνα έχει αποκλίνει από τις ειδικέ συστάσεις για, την ίδια, για τον εαυτό της. Άρα λοιπόν η κάθε χώρα αποφασίζει για το τι θα εφαρμόσει και τι όχι. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Διαφορετικά ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε η κάθε χώρα να δίνει θετικό input προς την Κομισιόν για τις γενικές συστάσεις προς την Ευρωζώνη και τις χώρες. Θα έπρεπε να είναι μια κυκλική και δημοκρατική προσέγγιση όπου οι συστάσεις δεν έρχονται απλώς εκ των άνω, αλλά είναι καρπός μιας ε, πραγματικής δημοκρατικής διαδικασίας συζήτησης με τα Εθνικά και το Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να αισθανόμαστε όλοι ότι οικειοποιούμεθα αυτήν την ε, διαδικασία του εξάμεινου και μάλιστα αυτή η έκθεση η Ροζάτη θα παίξει κρίσιμο ρόλο. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στον εντοπισμό, τρόπων με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε τη δημοκρατική διάσταση αυτού των εξαμηνίων κύκλων και από τις δύο πλευρές του κύκλου. με τρόπο ώστε να συμφωνήσουμε πώς θα τροφοδοτήσουμε την Κομισιόν από τη μια πλευρά και έπειτα να συζητήσουμε τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξει η Κομισιόν όσον αφορά την ετήσια έκθεση ανάπτυξη, τι γενικέ συστάσει για την Ευρωζώνη και τι ειδικέ για τα κράτη-μέλη. Και βεβαίω, λαμβάνοντα υπόψη τα όσα λέει το Κοινοβούλιο, στον τομέα μεταρρύθμιση τη διαδικασία και όχι μόνο ευθυγράμμιση, streamlining, έχουμε της, ε, τη σύγκληση των κατευθυντηρίων γραμμών όπου έχουμε καλύτερο ε, εντοπισμό στόχων και περισσότερο χώρο ελιγμού για τα κράτη-μέλη και για τα εθνικά κοινοβούλια που πρέπει να αποφασίσουν τα εφαρμοστικά μέτρα. Αυτή είναι το μίσο που μπορούμε λοιπόν να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε μαζί και πιστεύω επίσης πως το τομέα της ευθυγράμμισης του εξαμήνου θα ήταν πολύ θετικό να συζητήσουμε και να βρούμε έναν τρόπο ώστε να φτιάξουμε μια δημοκρατική συχνότητα για να ανταποκριθούμε και στη δημοκρατική ποιότητα και πιστεύω και στη ποιότητα της οικονομικής πολιτικής αυτού του εξαμήνου και της σχετικής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη συμβολή σας λοιπόν για αυτή, σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο μπορούμε. Δαρία, να λαμβάνουμε υπόψη το η συμβολή σας στην τελική μας έκθεση τόσο περισσότερο θα αυτή η χρονιά αυτή αυτή η συνεδρίαση εδώ θα συμβάλλει στις ευρύτερε μεταρρυθμίσεις της διαδικασία του εξαμήνου και στη διακυβέρνηση της ΟΝΕ. Είμαι βέβαιος πως ο εισηγητής θα βρει έναν τρόπο να έχει περισσότερο άμεση ε, άμεσο feedback σε συγκεκριμένε παραγράφου με βάση τις δικές σας προτάσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή συζήτηση και έτσι ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια μας διάταξη. Σας ευχαριστώ όλους. Τρία, λεπτά διάλειμμα για να ξαναφτιάξουμε τα έδρανα. Πάνω κάτω είμαστε στην ώρα μας.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 Okay. I, I sorry, I, we need to start our next point, which... Πρέπει να ξεκινήσουμε το εξέταση του επόμενου μας θέματος που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω όσους ε, πρέπει να φύγουν για όσους συζητούν, να συζητήσουν και να συνεχίσουν τη συζήτηση εκτός της αίθουσας. Λοιπόν, λοιπόν, μπορείτε να μείνετε αν θέλετε, είστε πρόσδεκτοι αν θέλετε να μείνετε και να ακούσετε και την συζήτηση αυτή για την έκθεση μπας, γιατί είναι σχετική με τα θέματα που συζητήσαμε. Δεν λέω λοιπόν ότι πρέπει να φύγετε, απλά κάντε ησυχία για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. μία 14 της ημερήσιας διάταξης. Απογραφή και προκλήσεις του νέου κανονισμού δημοσιονομικών ε, υπηρεσιών, αντίκτυπος και μελλοντικές κινήσεις για την Ένωση Κεφαλαγορών. Πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας να συμμετέχει ενεργά στη στρατηγική συζήτηση για την ε, ένωση των κεφαλογορών, τον αντίκτυπο κτλ. Πολύ σημαντικό λοιπόν να τροφοδοτήσουμε με την γνώμη μας ε, την Επιτροπή με έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Ε, τώρα λάβαμε το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή Μπούχερ Μπάλτσα και του δίνω αμέσω το λόγο για να μας την παρουσιάσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο έκθεσης ανταποκρίνεται σε μια απέτηση της Επιτροπής μας απέναντι στην Κομισιόν να εξετάσει δηλαδή την επίδραση της νομοθεσίας και όχι μόνο εξάντε άντε, εκ των προτέρων δηλαδή, αλλά και εξ Τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να περάσουμε νομοθεσία υπό πίεση χρόνου και έτσι συγκεντρώσαμε νομίζω κάποιες εμπειρίες ε, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν τώρα με το πέρασμα του χρόνου και ειδικά όταν ε, μιλάμε για νέες ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες γιατί οι στόχοι της Ένωσης των χρηματαγορών, δηλαδή να έχουμε τις βάσεις για μια σταθερή ανάπτυξη, θα επιτευχθούν μόνο εάν κοιτάξουμε όλους ε, τους ε, τομείς της, ε, των χρηματαγορών. Γνωρίζουμε πως συμμετέχοντας στην αγορά προέρχονται από διάφορους τομείς και βεβαίω ε, δεν μπορούμε να έχουμε μία ενιαία λύση για όλους γιατί υπάρχουν διαφορές ε, στο μέγεθο, στην πολυπλοκότητα και στο επιχειρηματικό μοντέλο και γνωρίζουμε πως η συνοχή και η συνέπεια στην ε, νομοθεσία δεν ήταν πάντα προτεραιότητα και άρα πρέπει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις για μία άρα σωστή ανάλυση δεν αρκεί μόνο να κοιτάξουμε τη χή, την ψηοδηγία ή κανονισμό, πρέπει να γίνει μια συνολική κοιταξουμε τη χη την ψιοδηγία η κανονισμο όλων των κλάδων των χρηματαγορών και να δούμε τι επίδραση θα έχουν στην πραγματική οικονομία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε πάρα πολύ για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και δικαίως η διαπίστωση πως συχνά λείπει η χρηματοδότηση ακούγεται από όλα τα στόματα όμως το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε η διαθεσιμότητα λύσεων που βασίζεται στις ε, κεφαλαιαγορές νομίζω είναι το πρώτο το οποίο σκεφτόμαστε όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν και διάβλη χρηματοδότησης άρα θεωρούμε πως και εδώ πέρα πρέπει να είναι συνολική και σφαιρική προσέγγιση και επιπλέον θα πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα κατά πόσον το ρυθμιστικό πλαίσιο ανταποκρίνεται στις ανάγκε των επενδυτών. Τα εμπόδια για διασυνοριακή πρόσβαση σε επενδύσεις ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ ψηλά. Η εσωτερική αγορά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, υπάρχει ήδη αλλά για τον καταναλωτή και τον επενδυτή δεν έχει υλοποιηθεί. Γι' αυτό προτείνω να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την ευρωπαϊκή προοπτική αλλά να κοιτάξουμε και, και να σκεφτούμε εκτός πλαισίου. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή και το διεθνές πλαίσιο, την διεθνή κατάσταση η οποία θα μας επηρεάζει όλο και περισσότερο. Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα άρα της Ευρώπης πρέπει να μας απασχολεί. Από την πλευρά του Αρμοδίου Επιτρόπου υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις πως είναι υπέρ μια συνολικής αξιολόγησης και σε σωρευτική βάση. Και αυτό βεβαίως ε, ταιριάζει και με την καλύτερη ρύθμιση και νομοθεσία που ζητάει η Κομισιόν. Βεβαίω υπάρχει ένα πολυεπίπεδο σύστημα. Καθώς ε, η πολυπλοκότητα του συστήματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι υπάρχουν ε, μεγάλες απαιτήσεις και από πλευράς αναλογικότητας και συνοχής. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε καλύτερα το χρονοδιάγραμμα και να βελτιωθεί η συνεργασία στην ομοθετική διαδικασία η Κομισιόν και οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία και στην εφαρμογή των νόμων. Νομίζω πως η Επιτροπή μας έχει δικαίωμα να εμπλακεί και στις δύο αυτές φάσεις. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως ανάβουμε κάποιο κόκκινο φως όσον αφορά την νομοθεσία. Πρέπει να πληρωθούν κάποιοι φάκελοι που αφορούν πράξεις κάτω εξουσιοδότηση και άλλες ε, προδιαγραφές. Γι' αυτό προτείνω να υποχρεώσουμε την Κομισιόν μέχρι τα τέλη του επομένου έτους να υποβάλει μια σχετική έκθεση και πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια των χρηματαγορών. Όπως ε, έγινε ήδη στο παρελθόν. Πρόκειται λοιπόν για κάποιε επιτυχίε οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν. Και τέλο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία για την βοήθεια στη σύνταξη του σχεδίου έκθεση και βεβαίω αναμένω τώρα την συζήτηση και την συνεργασία με τους σκιώδει συζητητέ. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα πρώτος ομιλητής είναι ο σκιώδης των σοσιαλιστών, ο κύριος Τάγκα. Πέντε λεπτά έχετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα ε, έκθεση ιδιαίτερα σε αυτή τη ε, διαδικασία ε, νομοθετικού έργου. Πολύ συχνά ε, είναι καλό εδώ να μπορούμε να ε, κάνουμε μια διαπίστωση, να κάνουμε μια απογραφή, ώστε να δούμε ε, ακριβώς πού βρισκόμαστε και πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. θα έπρεπε κανείς ε, να μπορεί να πει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι καλός, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο δημοσιονομικός τομέας ή δεν λειτουργεί. Εμείς θα θέλαμε ο δημοσιονομικός τομέας, ο χρηματοπιστωτικός τομέας να εξυπηρετεί την οικονομία. Αυτό είναι στο συμφέρον, προς το συμφέρον όλων και είναι δύσκολο να διατηρηθεί ένας τέτοιος χρηματοπιστωτικός τομέας γενικά ε, και να λειτουργεί προς όφελος όλων βλέπουμε σημαντικές ανισότητες. Ανισότητες ανάμεσα στις εταιρείε δεν είναι το ίδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για τους πολυεθνικούς ομίλους. Βλέπουμε ανισότητες ανάμεσα στις τράπεζες και αυτό έχει συζητηθεί ανάμεσα στις μικρές και μεγάλες τράπεζες αλλά και στις τράπεζες που εδράζουν σε διάφορες χώρες. Και έχουμε δει επίσης διαφορές στο είδος κεφαλαίου. Ας πούμε το ε, επισφαλές κεφάλαιο, ε, χρεόγραφα έναντι ε, χρέους και ούτω καθεξής. Ε, Επίση υπάρχει ανισότητα στην αντοχή στα οικονομικά σοκ και εξαρτάται από τα δάνεια και την ισχύ των στοιχείων, του ενεργητικού για να μπορέσουν να αντέξουν στα σοκ, στις εντάσεις. Και πάλι, όταν δει κανεί την ευρωπαϊκή αγορά, ε, μιλώ ευρύτερα, τράπεζε ε, μέχρι κεφαλαγορέ, βλέπουμε κατακαιρματισμό να επικρατεί. Και πραγματικά πρέπει να αναπτύξουμε από αυτό το πράγμα μια ατζέντα, όπως έχουμε ένα θεματολόγιο, όπως έχουμε κάνει και παλιότερα. Ε, ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση μάλιστα πριν το καλοκαίρι και πρέπει να τη συνεχίσουμε ώστε να καταλήξουμε σε ένα θεματολόγιο για να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε τις ανισότητες και με αυτόν τον τρόπο ο χρηματοπιστωτικός τομέας να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους περισσότερους, πραγματική οικονομία, τον κόσμο, τις επιχειρήσεις ε, προς τον οποίο το συμφέρον θέλουμε να ε, σκεφτόμαστε. Πολλά υποσχόμενες ενδιαφέρουσες επιλογές, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες, ε, που χρειάζονται ε, ιδιαίτερη προσοχή. Βλέπουμε, ας πούμε, τη δυνατότητα τυποποίησης της πληροφόρησης. Ας πούμε, ένα απλοποιημένο τρόπο, ένα πίνακα επιδόσεων, ε, ώστε να μπορεί κανείς πιο εύκολα να έχει πρόσβαση στις πιστώσεις, ε, αλλά και ολοκλήρωση του, της Ένωσης της Τραπεζικής. Υπάρχουν ακόμα πολλές διαφορές ανάμεσα στις τράπεζες και είναι σημαντικό να εκριζωθούν αυτές οι ανισότητες και επίσης θα πρέπει να επιταχύνουμε όχι με ένα βήμα τη φορά αλλά με δύο φορές όπως ας πούμε με το πλάνο ε, ασφάλισης των καταθέσεων. Ε, ταυτόχρονα δεν μπορεί να ξεχνάμε τα διδάγματα που καμίσαμε από τα τελευταία χρόνια. Ε, ε, πρέπει να δούμε, τη δυνατότητα ενός αποθετηρίου στοιχείων ε, που μας επιτρέπει εμάς τους, στους ρυθμιστές, τους επόπτες να εξετάζουμε τον χρηματοπιστικό τομέα, να βλέπουμε δηλαδή ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διατρέχουμε, σε ποιου κινδύνου εκτίθεται η πραγματική οικονομία λόγω αυτού του χρηματοπιστωτικού τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα χρεόγραφα ε, είδαμε ότι είναι πολύ προβληματική και περίπλοκη η κατάσταση. Πολλές φορές νομίζουμε πως είναι τελείως ανέφικτο να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν και κάποιες απλές... Ε, ευχαριστώ πολύ. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ε, τελείωσε ο χρόνος σας. Και του Σουίνμπορνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ε, εισηγητή για την εξαίρετη έκθεση γιατί εστιάζει στο μίσο που πρέπει να εξετάσουμε ώστε να μπορέσουμε να τελειοποιήσουμε τους κανονισμούς που συμφωνήθηκαν τα, τα περασμένα χρόνια και οι τομεί επί των οποίων θα επικεντρώσω τις τροπολογίες μου δεν θα εκπλέξουν τον εισηγητή γιατί αφορούν ε, την, το το οποίο ε, και μετά έχω τρία ευρύτερα θέματα τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Είναι τομεί που θα πρέπει να εξετάσουμε. Ε, νομίζω σε αυτό συμφωνεί και ο εισηγητής. Είναι η αναλογικότητα για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Ε, το η προσοχή που πρέπει να δώσουμε στη ΣΕΖΑ και ε, τα αντίστοιχα καθεστώτα στις ε, ε, τρίτες χώρες. Ας πούμε στο ΕΜΙΡ μπορούμε να κάνουμε πολύ, σε πολλά πράγματα όπως η τυποποίηση της αναφοράς. Είχε γίνει η δουλειά το 2000 2010, αλλά δεν είχαμε πολλέ τροπολογίε ούτε πολλέ αντιφάσεις και υποτίθεται ότι ήταν απλό το ζήτημα. Όμως στην πράξη δεν ήταν τόσο απλό τελικά. Ε, καθώς έθιξε αυτό το θέμα υπάρχουν τουλάχιστον 89 ε, διαφορετικοί ε, τομείς αναφοράς υπό το ΕΜΗΡ και δεν ευθυγραμμίζονται με, την, με τις αναφορές του CFDC ούτε οποιοδήποτε άλλου διεθνούς οργανισμού. Ε, τελικά οι δημοσιονομικοί υπόπτες θα έπρεπε να βλέπουν, να μπορούν να δουν ποια είναι η διασύνδεση ανάμεσα στους διεθνείς παίκτες. Γιατί όταν είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δεν μπορεί κανείς να το εξετάσει, ε, τότε δεν εξυπηρετεί το σκοπό που, για τον οποίο το φτιάξαμε. Για να παραθέσω τα σχόλια του Λουξεμβούργιου Υπουργού Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα, φτιάχνουμε ένα τεράστιο πολλό νεκροταφείο από διάφορα στις νομοθεσίες. Ε, θα πρέπει να όλα αυτά λειτουργούν μόνο όταν ομοιόμορφα το εφαρμόζουμε χωρίς να περιπλέκουμε τα πράγματα με ιδιαιτερότητες εξωπεριφερειακές. Αυτό σημαίνει ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να ηγηθεί ε, σε αυτό το θέμα. Ε, άλλο βασικό στοιχείο είναι ε, ότι πρέπει να απλοποιήσουμε την αντιμετώπιση των μη χρηματοπιστωτικών ε, συμβαλόμενων μερών, γιατί οι εθνικοί εμπειρογνώμονε βρίσκουν ορισμένε στοιχείε πολύ δύσκολε στην εφαρμογή του και στην ερμηνεία του, πράγμα που δεν βοηθάει τι εταιρείε ούτε του επόπτε ολόκληρη την Ένωση. Και αυτό είναι και το κεντρικό σημείο που ανέφερε ήδη ο κ. Μπόλ στην εκθεσή του όσον αφορά άλλου τομεί νομοθεσία. Η Ένωση Κεφαλαγορών θα πρέπει να εξετάσει μόνο τα μεγάλα προγράμματα όπως η τιτλοποίηση, αλλά και να προσθέσει μικρά ε, κόλπα ή επιλογές, ε, options που υπάρχουν στις ισχύοντες κανονισμούς, έτσι ώστε οι μικρομεσαίες τράπεζες ε, να μπορούν να συμμετέχουν και να αντιμετωπίζουν τις διάφορες ανάγκες των ίδιων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως και κάποια πρακτικά παραδείγματα επιβολής ε, των θέσεών τους στους τριμερείς διαλόγους. Τα παραδείγματα για τις ομίλους ή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να είναι παραθυράκια εφόσον υπάρχει κατάλληλη εποπτεία. Και νομίζω ότι το να μην επιτραπούν παραθυράκια στο προηγούμενη θητεία και αυτή η αγωνία οδήγησε σε πολύ άκαμπτους κανόνες. Τώρα, για την λειτουργία των ΕΣΑ. Ε, ανησυχώ για τις διαφορετικές προσεγγίσεις ε, σχεδιασμού των κανόνων επίπεδου 2 όταν πάμε προς την Κομισιόν και πόσο σκληρά πρέπει να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε την επικοινωνία με το Κοινοβούλιο σε τομείς όπως η Δεδομένου ότι οι κανόνες επίπεδου 2 υιοθετούνται ε, με βάση το 2.19 και το και το 2.91 θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει συνεργασία. Η Κομισιόν συζητά τα σχόλια που εμείς στέλνουμε με τους εθνικούς πυρογνώμονες και μετά έχουμε διάφορα στάδια ανάπτυξης όλων αυτών. Έχουμε δύο στάδια συντάξεις αλλά όταν φτάσουμε στην RTS, ας πούμε, δεν πήραμε κανένα σχέδιο από την ΕΣΜΑ. Και μόνο και τμήμα της διαπραγματευτικής ομάδας. Και πολύ φοβάμαι ε, για τις ε, δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να μας περιμένουν όταν θα φτάσουμε στην ε, πραγματική διαπραγμάτευση. Και για τις φήμες που μπορεί να μας ενδιαφέρουν, αυτό δεν εμποδίζει τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Προσαρμογές και καθυστερήσεις είναι βλαβερές ε, για την πρόοδο των ΕΣΑ και δεν είναι κάτι που και εμείς επιθυμούμε. Δεύτερη μου παρατήρηση αφορά πάλι τη ΕΣΑ και αφορά το ενιαίο εγχειρίδιο και την προσέγγιση αυτή και πώς αυτή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Θα ήθελα να δω πώς ο μηχανισμός παρακολούθησης των, ετε, των εταίρων μπορεί να οδηγήσει στην ποιότητα της εποπτείας. Διακόπτει ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την ύπαρξη της έκθεσης αυτής που είναι ε, ισορροπημένη και ολοκληρωμένη, περιεκτική. Χαίρομαι διότι δίδεται έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε, κάθε αθρηστική αξιολόγηση θα πρέπει να ε, ε, αξιολογεί και ζητήματα όπως είναι η πρόσβαση των ΜΜΕ μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Θεωρώ ότι ε, τα αναπτύσσονται οι αγορές, υπάρχουν οι αναδυόμενες αγορές, αναπτυσσόμενες αγορές στην Ασία και πρέπει να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση της νομοθεσίας ε, για τα χρηματοπιστωτικά. Πρέπει να ευθυγραμμιστεί η σχετική νομοθεσία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να είναι ηγέτης στην παγκόσμια αγορά χρηματοπιστωτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Χαίρομαι διότι στις παραγράφους 24 και 25 γίνεται αναφορά στο θέμα των ισοδυνάμων και των αντιστοιχειών και θα πρέπει αυτά να γίνονται με συνέπεια. σε σχέση με την επιστολή που στείλαμε στον Επίτροπο Χίλ. Ο Επίτροπος είπε ότι είναι δύσκολο να καθοριστούν ε, κριτήρια για την αντιστοιχία ή την ισοδυναμία γιατί ε, ε, κάθε μέτρο εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό. Όμως πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω τους σκοπούς της εναρμόνισης των πλαισίων ισοδυναμίας ή αντιστοιχίας και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πράξει. Ε, χαίρομαι γιατί θέλω πολύ να συνεργαστώ και με τον εισηγητή και με τους χιώδες εισηγητές της επόμενης εβδομάδας και ελπίζω η έκθεση να εγκριθεί. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος ευχαριστώ, Φάμπιο Ντεμάση. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για την έκθεση. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θα μείνω για όλη τη συζήτηση. Έχω δυστυχώς και άλλες ε, δουλειές πρέπει να κάνω γαλλικαρισμό της ομάδας. θα ήθελα να πω πως ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάποια πράγματα, δηλαδή να δούμε ποιοι είναι, ποια είναι η φυστάμενη κατάσταση, αλλά θεωρούμε πως είναι σημαντικό να δούμε τα κενά όσον αφορά την ρύθμιση των ε, χρηματαγορών και όχι με τη λογική να δούμε τι μπορούμε να ξεφορτωθούμε. Δεύτερον, θεωρούμε πως είναι σωστό αυτό το οποίο λέμε πως υπάρχουν άλλοι επικαλύψεις, υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα, αλλά βασικό πρόβλημα της ρύθμισης αυτού τομέα είναι πως είναι πολύ πολύπλοκες οι ίδιες οι χρηματαγορές και μια σωστή ρυθμισή θα μείωνε αυτή την πολυπλοκότητα και θα πρέπει να δώσουμε βέβαια προτεραιότητα στην σταθερότητα και βλέπουμε επίσης τεράστιο κίνδυνο εδώ πέρα. Τώρα, το ποιο θα είναι το κόστος εάν δεν εστιάσουμε σε αυτή την ε, σταθερότητα είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, ένας ε, προσανατολισμός προς τα εκεί, γιατί βεβαίως έτσι θα δούμε ότι το κόστος της γραφειοκρατίας είναι μηδαμινό μπροστά σε αυτό. Επίσης, μέχρι στιγμής η ρύθμιση των χρηματαγορών προσανατολιζόταν στον ε, μικρο τομέα, δηλαδή κοιτάγαμε ισολογισμούς κτλ. Αλλά στο, στο μάκρο επίπεδο δεν κοιτούσαμε αρκετά συστημικούς κινδύνους Και, τα λοιπά. και όταν μιλάμε επίσης για μια Ένωση αγορών ιδιαίτερα. Σας είπα, εμείς είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και οι κεφαλαιαγορές ε, είναι κάτι το συμπληρωματικό. Στην Ευρώπη έχουμε ένα τραπεζοκεντρικό σύστημα το οποίο έχει πλέον εκτίματα για την ε, ασφαλή χρηματοδότηση. Το τωρινό πρόβλημα τώρα εμείς θεωρούμε ότι δεν οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης. Υπήρξε ένα άρθρο πριν από λίγες μέρες του Lord Simmons στην ε, Financial Times και είπε πως το πρόβλημα είναι ο χαμηλός τζίρος, όχι η έλλειψη χρηματοδότησης. Οπότε θεωρούμε πως το καλύτερο μέσο για να κινήσουμε την πίστη και τις επενδύσεις είναι να σταθεροποιηθεί η ζήτηση και ο όρος αυτός που εμφανίζεται συχνά, η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα γιατί η ανταγωνιστικότητα ε, συχνά την μεταφράζουμε σε μέγεθος. Αυτό δεν είναι αυτός σκοπός, ειδικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ε, επιχειρήσεων. Ένα αποκεντρωμένο σύστημα είναι πολύ πιο επιτυχημένο. Έχουμε τα διάφορα τοπικά ταμιευτήρια στη Γερμανία που βγήκαν σχετικώ αλόβητα από την κρίση. Και τέλος επίσης να επισημάνω θετικά πω υπάρχει μια πτυχή που με έπεισε λέει ο κύριος Μπούκχατ εδώ πέρα πρέπει να δούμε την διάκριση μεταξύ πράξεων κατεξιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων δεν πρέπει να μας πάρουν εδώ πέρα την νομοθεσία μέσα από τα χέρια και οπωσδήποτε το στηρίζουμε αυτό 100% ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Μπορκ για την έκθεσή του. Ε, υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία συμφωνούμε. Πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να δούμε το θέμα της αναλογικότητας και να ελέγξουμε την νομοθεσία. Βλέπουμε πάρα πολλές ε, συνέπειες ε, οι οποίες είναι μη σκεμμένες ακούσιες συνέπειες της νομοθεσίας μας και της ρυθμισής μας οπότε χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα θα έλεγα ναι. καθώς ε, θα πρέπει να δούμε εάν και στην ε, νομοθεσία υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία θα καθορίζουν την αναλογική συμπεριφορά των εποπτικών αρχών. Επίσης, αυτό το οποίο λέγεται ως ε, relationship banking και το εάν λαμβάνει σωστά την αρχή ίδιες αρχές για ίδιους κινδύνους και ίδιοι κανόνες για όλους. Πρέπει να δούμε εδώ πέρα πώς θα τηρηθούν και τα δημοκρατικά μας ε, δικαιώματα. Γιατί κάπου έχουν ξεφύγει τα πράγματα και πρέπει να τα δούμε. Οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε την έκθεση αυτή και το θέμα είναι εδώ πέρα και εδώ συμφωνώ με τους σοσιαλιστές ότι καταφέραμε το σύστημα σήμερα να εξυπηρετεί περισσότερο την πραγματική οικονομία από ό,τι στο παρελθόν και να πηγαίνει και μεγαλύτερο μέρος των κερδών στον επενδυτή αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι μια κατασκευή μπαρόκ, πάρα πολύ ακριβή και εις βάρος και της πραγματικής οικονομίας και των επενδυτών. Πρέπει να έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο θα υπηρετεί την πραγματική οικονομία και θα προσφέρει και αποδόσεις στους ε, επενδυτές και δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ε, όπου οι αποδόσεις ε, θα καταλήγουν σε πανάκριβους ε, πύργους τραπεζιτών αντί να πηγαίνουν σε αυτούς οι οποίοι επενδύουν τα λεφτά τους. Επίσης θεωρούμε πως η νομοθεσία έχει γίνει κάπου υπερβολικά περίπλοκη και λέτε πως θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις για το πως θα μπορέσουμε να φέρουμε μία τάξη στην ε, κατάσταση αυτή. Θεωρώ πως θα πρέπει πράγματι να γίνει αυτή η συζήτηση, η οποία είχε γίνει και στο στην προηγούμενη θητεία. Έχουμε το θέμα των σκιωδών τραπεζών και της σκιώδους ε, τραπεζικής. Πρόκειται λοιπόν για επιχειρήσεις που έχουν ένα παρόμοιο προφίλ κινδύνου, αλλά ε, έχουν διαφορετικούς κανόνες και το ερώτημα είναι τι έχει κάνει η Κομισιόν εδώ πέρα σε επίπεδο G20 και FSB. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε πως ε, η εσωτερική αγορά έχει κάπως εμβαθυνθεί αλλά έχουμε πάρα πολλές εξαιρέσεις κάποιες από τις οποίες είναι αιτιολογημένες, άλλες όμως όχι. Τα ανέφερε τα προβλήματα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και νομίζω πως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά για να μπορέσουμε ακριβώς να λειτουργήσουμε με το κοινό νόμισμα. Τέλος, υπάρχει μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης στην αγορά. Έχουμε τις ε, υπηρεσίες και τους οίκους αξιολόγησης Προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται άρα με τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και την ισχύ που τους δίνει αυτό. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Θέλουμε παντού ένα πραγματικό ανταγωνισμό. Πάρα πολλούς ε, παίκτες ε, και εδώ πέρα δεν έχει σημειωθεί η πρόοδος. Και τέλος, κάτι το σημαντικό για εμάς, ότι θέλουμε Βεβαίω, βιώσιμες επενδύσεις, να υπάρχει ένα οικολογικό και κοινωνικό πρόσημο, το κεφάλαιο να πηγαίνει στους κατάλληλους τομείς που θα ωφελήσουν το μέλλον και βεβαίως ε, να στέλνει τα σωστά μηνύματα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για την συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Στίβεν Κούλφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την πράσινη βίβλο που αναφέρει, αναφέρεται στην δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών αναφέρεται η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, που είναι να έχουμε θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας τρόπος είναι να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στις ευρωπαϊκές υποδόμες. Συμφωνώ απολύτως. Ενισχύουμε τις ε, επενδύσεις έχοντας μία ένωση κεφαλαγορών και έτσι βελτιώνουμε τα κεφάλαια που δίδονται. Αναφέρεται ότι τα εμπόδια για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης αγοράς κεφαλαγορών είναι οι κατακαιρματισμένες αγορές, τα εμπόδια στο εσωτερικό της κάθε αγοράς, κυρίως χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από πλευράς προσφοράς οι αποταμιεύσεις δεν πηγαίνουν μέσα στο σύστημα στο βαθμό και με τη ταχύτητα που θα θέλαμε. Και λέγεται επίσης ότι αξίζει να έχουμε μια ένωση κεφαλαγορών, διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους δέχονται πέντε φορές περισσότερη χρηματοδότηση από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λέγονται. Εγώ τις ε, διάβασα αυτές τις εκθέσεις και θέλω να επαναλάβω το αρχικό μου σχόλιο. Φαίνεται σαν να είναι ένα εγχειρίδιο για τους μη μοιημένους στις ε, χρηματαγορές και στις κεφαλαγορές. Ίσως ε, είμαι νεοφώτιστος και δεν ε, γνωρίζω πολλά. Θέλω όμως να τονίσω τις τεχνικές πτυχές αλλά κυρίως την προσέγγιση που ακολουθείτε. Καταρχάς η σύγκριση με τη ΣΥΠΑ είναι ένα ελάττωμα σχεδιαστικό που προσπαθεί αυτό το μέρος να αντιγράψει. Καταρχάς η Ευρώπη απαρτίζεται από πολλές και λαμπρές χώρες και από πολλούς και λαμπρούς λαούς. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι μία χώρα με μία σειρά κανόνων και ένα μόνο λαό. Και τον Αμερικανικό λαό. Και πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Είναι ένα θεμελιωδές ε, φιλοσοφικό ζήτημα το οποίο δεν εξετάζεται σε αυτή την έκθεση. Δεύτερον, η λύση που προτείνεται δεν θα βοηθήσει πάντοτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως περιμένετε εσείς. Πράγματι, μπορούν να πάνε στις τράπεζες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη και να πετύχουν αρκετά. Όμως, ο τραπεζικός κλάδος δεν επενδύει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όχι γιατί δεν αξίζουν αυτές απαραίτητος, αλλά διότι ο κίνδυνος τους το απαγορεύει και ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας φαίνεται αρκετά σκιώδης και δεν λύνονται αυτά τα ζητήματα με την απλή επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγορών, αγορών κεφαλαίου κτλ. Από εκεί και πέρα οι μυρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν διάφορες δυσκολίες και θέλω να παραθέσω τον επικεφαλής της Γερμανικής Ένωσης ε, Αποταμευτικών Τραπεζών, ο οποίος λέει ότι το κόστος της παραδοσιακής τραπεζικής ε, ε, θα είναι πολύ μεγάλο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να πετύχουν ανάπτυξη γιατί εταιρικά ομόλογα αξίας κάτω των 10 εκατομμυρίων θα είναι ομόλογα στα οποία δεν θα αξίζει πάρα πολλοί θεσμικοί επενδυτές να επενδύσουν οι οποίοι ε, δεν ενδιαφέρονται αν έχουμε νούμερα κάτω των 25 εκατομμυρίων, δηλαδή ομόλογα. Άρα υπάρχει ήδη αυτός ο διαχωρισμός και πρέπει συνεχώς να είναι όλο και πιο αυξημένα τα εισιτήρια ε, για να πάρει κανείς το εισιτήριο εισόδου και να τραβήξει επενδυτές. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας που μιλά ε, για τα εμπόδια της επένδυσης των οικοκυριών στις κεφαλαγορές. Δηλαδή θέλουμε να θαρρύνουμε τα νοικοκυριά να μην αποταμιεύουν τις αποτιμήσεις τους στις τράπεζες, κάτι το οποίο είναι και το πιο ασφαλές εκτός και αν είναι κανείς Κύπριος όπου εκεί την είχε πολύ δύσκολα. Θέλουμε τα νοικοκυριά να επενδύουν τις αποτεμιεύσεις τους στις τιτλοποιήσεις. Μα από τις τιτλοποιήσεις χάσαν πάρα πολύ χρήματα κατά τη διάρκεια της κρίσης και του κράχ. Και Έχουμε περιορισμού στα ίδια κεφάλαια γιατί αυξήνουμε το κόστος κεφαλαίου, τα προαπαιτούμενα, τα, τις κανονιστικές ρυθμίσεις και θέλουμε να και αυτά εμποδίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επενδύσουν ή να χρηματοδοτηθούν και από την άλλη ενθαρρύνουμε τα νοικοκυριά να μπουν ε, σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου για το έγγραφο ε, αυτό. Ευχαριστώ. Η Μπάρμπαρα Κάπελ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πίσω από αυτό το μεγάλο τίτλο της έκθεσης ε, κρύβεται μια σημαντική έκθεση για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. και αφορά τον έλεγχο εξ και εξ της ε, νομοθεσίας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα και είναι σημαντικό το το κάνει αυτό ο εισηγητής του ΕΛΚ γιατί η έκθεση έχει πολύ μεγάλη σημασία. το πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα το δείχνουν ε, τα επόμενα βήματα που υπάρχουν στο σχέδιο έκθεσης τα οποία στηρίζω δηλαδή ετήσια επανεξέταση της ε, συνοχής και της αναλογικότητας ειδικά όταν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και πενταετής ποσοτική και ποιοτική εξέταση των επιπτώσεων. Σημαντική είναι, όπως είπαμε λοιπόν, και η χρονική αυτή πτυχή, ότι η Κομισιόν μέχρι το τέλος του επομένου έτους δηλαδή θα πρέπει να υποβάλει μια έκθεση αντικτύπου, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να εξεταστούν ε, όλοι οι κλάδοι των χρηματαγορών, αναφέρθηκε πολλές φορές, είναι περίπλοκος ο τομέας, αδιαφανής, αλλά είναι σημαντική η εξέταση, γιατί βεβαίως πρέπει να εξεταστεί και η πραγματική οικονομία και ήδη είπαν οι προλαλήσαντες πως εάν συγκρίνουμε ε, με τις ΕΠΑ, στις ΕΠΑ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν πέντε φορές περισσότερα κεφάλαια από τις ε, χρηματαγορές σε σχέση με την Ευρώπη στο χρονικό διάστημα 2008 με 2014 όταν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, θα είχαν ε, αυτά τα 90 δισεκατομμύρια παραπάνω σε χρηματοδότηση που είχαν οι αμερικανικές ε, επιχειρήσεις αν τις συγκρίνουμε. Και ακριβώς αυτοί οι διάβλοι οι οποίοι δίνουν στην πραγματική οικονομία χρηματοδότηση πρέπει να εξεταστούν και να τονιστεί αυτό σε αυτή την έκθεση. Στόχος είναι να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε πιο στοχευμένα, όπως είπαμε, τους κανόνες με στόχο την προστασία του καταναλωτή, την σταθερότητα και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, η οποία βέβαια είναι σημαντική γιατί, υπόθηκε, τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε διεθνή ανταγωνισμό και στον διεθνή αυτόν ανταγωνισμό πρέπει να μπορούν να σταθούν. Αυτά είναι τα σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη και θεωρώ πως θα τύχει θετική υποδοχή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ε, τρεις που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις στη διαδικασία Catch the Eye. Ένα μισή λεπτό ο καθένα σας και η κάθε μία σας παρακαλώ, γιατί έχουμε ε, ξεφύγει από το χρόνο μας, έχουμε καθυστερήσει. Και δεν ξέρω ποιος μπορεί να με αντικαταστήσει στη συνέχεια, μάλλον κανείς και θα πρέπει να φύγω σε 6.30 γιατί έχω άλλη σύσκεψη. Η Νίνα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για την καλή του έκθεση και στηρίζω πολλά από τα συμπεράσματα στα οποία έχετε φτάσει και στηρίζω και αυτό που λέει ο συνάδελφος Τάγκα. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ των διαφόρων νομοθετημάτων για τα χρηματοοικονομικά και θα πρέπει αυτό να το δούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια αίσθηση διάχυτη και την έχω δει σε διάφορες συναντήσεις που έχω με ανθρώπους από το χρηματιστηριακό κλάδο. Πιστεύουν ότι το εγχείρημα που κάνουμε για την ε, καταγραφή της νομοθεσίας ε, ε, είναι ένα εγχείρημα για να ε, μειώσουμε την νομοθεσία. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μια διαδικασία απορρίθμισης, είναι μια διαδικασία λίανσης των δυσκολιών και τελειοποίησης και θα πρέπει αυτό το μήνυμα να το στείλουμε. Ο ετήσιος έλεγχος τώρα. Θέλω να καταλάβω περισσότερο πόσο εύκολο είναι και πόσο πρακτικό είναι να γίνεται κάτι τέτοιο. Και είναι μια ιδέα την οποία θα πρέπει να διερευνήσουμε παραπάνω. Ωστόσο, πράγματι χρειαζόμαστε πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση της νομοθεσίας που έχει ήδη υιοθετηθεί. Ε, θα πρέπει να μην ε, γυαλίζουμε μόνο τα ασημικά, αλλά να δούμε ε, τα πραγματικά προβλήματα για να έχουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφάλαια Αγορών. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κι εγώ. Ήθελα να πω στον κύριο Γούλφ ότι αν έρθει μία μέρα που ο Τζέρεμι Κόρμπιν εκλεγεί Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εκτό του Ηνωμένου Βασιλείου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πολύ θα νοσταλγήσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τι Χρηματαγορέ. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Ε, ε, αποτίμησε τη βάση στην οποία βρισκόμαστε και αυτό είναι σημαντικό. Θα ακολουθήσω λοιπόν τη γραμμή του και θα προσθέσω ότι καλό είναι να γίνει ανάλυση από τη μακροοικονομική σκοπιά. Έχουμε αντιμετωπίσει τις χρηματιστηριακές αγορές, χρήματα αγορές και χρηματοπιστωτικές αγορές με τρόπο ώστε να δίνουν τις επενδύσεις που χρειάζομαι στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί κανονισμοί που υιοθετήσαμε, καλό ή κακός, τελικά τους δυσκόλεψαν τη ζωή και το λέω ε, καλό ή κακός γιατί μερικές φορές ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υιοθετηθούν τέτοιου είδους νομοθεσίες και άλλες φορές ήταν εξαιρετικά εύκολο. Εν πάση περιπτώσει τους διευκολύναμε να επενδύσουν περισσότερο στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Καλό είναι να συζητήσουμε για το τι έχουμε πετύχει. Όλα ήταν καλά αυτά που πετύχαμε. Μήπως έκαναμε υπερβολικά πολλά ή μήπω κάτι δεν κάναμε και υστερούμε. Και η σταθερότητα των χρηματαγορών εξαρτάται από την ανάπτυξη ούτως ή άλλως και έχουμε πολύ εύρυθμα λειτουργούσες κεφαλαγορές ορισμένα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε αυτές ως παράδειγμα. Μόνο 5 δευτερόλεπτα ξεπέρασα τον χρόνο. Είναι πολύ χαμηλές οι επιδόσεις αυτές έτσι δεν είναι. Ο Πρόεδρος. Η αναλύση. Ναι, θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Χαίρομαι για την εμπιστοσύνη του κυρίου Χόκμαν, ο οποίος πιστεύει ότι το κόμμα μου θα ε, κερδίσει τις επόμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε, η Ένωση Κεφαλαγορών πράγματι είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι Βρετανικές επιχειρήσεις τείνουν να υποστηρίζουν την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όλα αυτά που λέγονται στην έκθεση και ευχαριστώ τον εισηγητή. Όταν όμως ο εισηγητής αναφέρει τις αρχές που θα πρέπει να μας διέπουν, ε, δεν έχει βάλει μια πολύ σημαντική, την αρχή της διαφάνειας και αυτό είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης όσων εμπλέκονται στις αγορές κεφαλαίου και την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού. Ελπίζω να τονίσει περισσότερο ε, την διαφάνεια, γιατί δεν την βλέπω πουθενά στην έκθεση. Αυτό καταρχάς. Δεύτερον, πολλή συζήτηση έχει γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις προοπτικές κανονιστικών αλλαγών, αλλαγών του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και το πιο ε, ε, συχνό σχόλιο των επενδυτών είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι ακόμα έτοιμες και χρειάζονται την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει και αυτά να τα δούμε και να τα εξηγήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εισηγητής κύριος Πάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ε, παρατηρήσεις τους θετικές ή αυτές που έλεγαν ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά. Μπορώ να σχολιάσω πολλά πράγματα, αλλά για λόγους χρόνου περιοριστώ σε λίγα βασικά. Το είπε ο κύριος Ντότζ, το θέμα της διαφάνειας. Πράγματι, Είμαι διατεθειμένος ε, να το ξαναδώ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έφυξαν το θέμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρώ πως ε, πρέπει να δώσουμε σημασία και σε αυτό. Πρέπει να δούμε το ζήτημα αυτό. Όπως είπε και ο Πέτριγέζικ είναι ένα σημείο κλειδί. Επίσης, συμφωνώ με τον Πολ Τάγκ ότι έχει πραγματικά φτάσει η ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό και αναφέρθηκε νομίζω ήδη ότι απαιτείται κάτι τέτοιο. Είναι η Τζιλ νομίζω ήταν αυτή η οποία είπε ότι πρέπει να κάνουμε μια ρύθμιση στις λεπτομέρειες και όχι κάποια απορρίθμιση. Δεν ανάβουμε κανένα κόκκινο φως, απλά θέλουμε να δούμε τι μπορεί να βελτιωθεί στην νομοθεσία των τελευταίων ετών. Κατά την άποψή μου, είναι επίσης σημαντικό να δούμε το ζήτημα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, το είπε και ο Φάμπιο Ντεμάζη. Είναι θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και πολύ μάλιστα και σύντομα για αυτό το οποίο είπε ο Σβέν Γίγκολτ. Ναι, ο έλεγχος αναλογικότητας είναι σημαντικό θέμα και επειδή όμως συνολικά η νομοθεσία είναι υπερβολικά περιπλοκή κάτι το οποίο με απασχολεί εμένα πάρα πολύ είναι αυτό το οποίο ανέφερες για την σκιώδη τραπεζική υπεσία, εγώ θα έλεγα σκιώδη οικονομία ολόκληρη. αλλά έχω την προσωπική πεποίθηση πως αυτό θα είναι από τα μεγάλα ζητήματα της εκλογικής περίοδου. Το τι θα κάνουμε δηλαδή με αυτά τα ζητήματα μια σύντομη παρατήρηση τώρα Δεν είπα πως ε, επειδή έκανα μια αναφορά στις ΗΠΑ δεν νοούσα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ομοσπονδιακό κράτος μην με παρεξηγήσετε ε, δεν είναι αυτό το θέμα της έκθεσης ούτως ή άλλως και ούτως ή άλλως ε, άλλες είναι οι επιτροπές που είναι αρμόδιες. Όσον αφορά λοιπόν τον ρυθμό της ε, επανεξέτασης, ε, ευχαριστώ να το συζητήσω με τους ηγητές, αλλά αποφάσισα εσκεμένα να κάνω αυτή την πρόταση γιατί θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο τέλος. Θεωρώ πως το μήνυμα εδώ πέρα στο τέλος θα πρέπει να είναι πως ε, χρειαζόμαστε καλή δουλειά, μια μελέτη των επιπτώσεων, ε, να μας κάνει μια καλή μελέτη επιπτώσεων κομισιών και να έχουμε ένα σαφές μήνυμα προς την κατεύθυνση της ε, κομισιών. Αυτά νομίζω είμαι κοντά στα 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Για να δω τα επόμενα βήματα. Έχουμε προθεσμία για υποβολή τροπολογιών στις 24 ε, Σεπτεμβρίου, εξέταση των τροπολογιών 13 Οκτωβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ στις 9 ή 10 Νοεμβρίου. Επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΟΝ θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα στη συνεδρίαση.